Καλησπέρα σας λοιπόν. Νομίζω ότι είναι ώρα να ξεκινήσουμε πλέον Έχουμε σαν πρώτο σημείο τη ημερησία διατάξεω μα σήμερα το απόγευμα ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο κ. Λάσλο Κόβαξ. Είμαι πάρα πολύ ευτυχή που μπορώ να δεχτώ τον Επίτροπο στην Επιτροπή. Πρέπει να σα πω ότι ήταν ο πρώτο Επίτροπο ο οποίο ήρθε άμεσα σε επαφή μαζί μου ε, και ε, αναφέρθηκε σε κάποια σημαντικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολήσουν και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό. Θα ήθελα να πω στους παρισταμένους ε, πώς θα ακολουθήσουμε, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ένα νεύμα και με την ε, κάρτα σας ε, και να ε, εγγραφείτε στον γύρο ερωτήσεων. Αφού λοιπόν κάνει την κεντρική του παρέμβαση ο Επίτροπος, τότε θα ξεκινήσουμε δίνοντας τον λόγο στον πρώτο αγορητή αναομάδα. Καλό θα ήταν να είναι και ο συντονιστής της ε, ομάδας. Και μετά θα δούμε catch the eye. Όποιος σηκώνει το χέρι του θα παίρνει τον λόγο. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε δηλαδή μια ανταλλαγή εξαιρετικά αυστηρή όπως θα ήταν ας πούμε με τον κύριο Τρισέ όπου θα δίνεται ο λόγος βάσει της αναλογικής δύναμης των ομάδων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο και νομίζω ότι χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα πρέπει να του δώσω το λόγο. Ε, και να του δώσω το λόγο για να μας πει οτιδήποτε προτίθεται και έχει διάθεση να μας πει. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Επίτροπος. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούν οι διερμηνείς, δυστυχώς. Before starting... Πριν ξεκινήσω την ε, ε, πραγματική μου αναφορά στα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, Νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο δημοψήφισμα της Ιρλανδίας, γιατί εκατομμύρια Ευρωπαίοι ή μάλλον δεκάδες εκατομμυρίων ε, είναι πάρα πολύ ευτυχής διότι επιτέλους το εκλογικό σώμα της Ιρλανδίας είπε το μεγάλο ναι στην συνθήκη της Λισαβόνας και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή η απόφαση του εκλογικού σώματος της Ιρλανδίας θα προωθήσει κατά μεγάλο μέρος τη διαδικασία κύρωσης, έστω και αν ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα ε, εκκρεμότητες ε, με δύο χώρες, με την Ολλανδία και με την ε, Τσεχική Δημοκρατία συγκεκριμένα. Πάντως πραγματικά ελπίζω ότι θα προχωρήσει η κύρωση της συνθήκης και από τις δύο αυτές χώρες όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όταν και εφόσον τεθεί σε ισχύ η ε, συνθήκη της Λισαβόνα θα έχουμε μεγαλύτερη δημοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σίγουρα καλύτερη λειτουργία του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επομένως αυτό θα είναι προς όφελος 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό ήθελα να σας πω γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ε, είμαι ιδιαίτερο ικανοποιημένος και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά και την ικανοποίησή μου για την έκβαση της πληροφορίας στην Ιρλανδία. Τώρα, ε, πλησιάζω στο τέλος της θητείας μου στην θέση του Επιτρόπου Αρμοδίου για τη Φορολογία και την Τελωνιακή Ένωση και θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την φιλοσοφία που έχω όσον αφορά την, ε, την ευρωπαϊκή ιδέα, αντίληψη για φορολογία. Πιστεύω ότι η φορολογία αυτή θα πρέπει να έχει μοναδικό στόχο την προώθηση της ενιαίας αγοράς και βεβαίως και την προώθηση της εφαρμογής των κεντρικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την ε, δυνατότητα επίτευξης των στόχων της να προωθήσει δηλαδή την ανάπτυξη, να στηρίξει τις πολιτικές ε, ε, απασχόλησης, να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κυρίως δε εδώ στα πλαίσια της κρίσης να διατηρήσει θέσεις εργασίας, να ε, διατηρήσει την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια όσον αφορά την ενέργεια, να να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων, των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας ξεκινήσω λοιπόν με κάτι που τώρα αποτελεί παρελθόν όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία, δηλαδή ε, τι, το θέμα του ε, ΦΠΑ και της αναθεώρησης του ΦΠΑ. Ε, πρόκειται για μία συζήτηση που κράτησε δέκα χρόνια. Ε, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ επέτυχε ε, συμφωνία όσον αφορά την διαρκή εφαρμογή τη εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ σε ειδικέ περιπτώσεις ε, για ασφάλεια, για συγγνώμη, περίθαλψη στο σπίτι, για ε, την εστίαση και σε περίπτωση μόνο κατά την οποία χρησιμοποιεί, ε, βρίσκεται σε τοπικό επίπεδο και χρησιμοποιεί και προϊόντα της τοπικής αγοράς. Διευρυμένη διευρυμένη ε, χρήση των μειωμένων ποσοστών του ΦΠΑ θα μπορούσε να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης και να σώσει ε, δεκάδες και εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά κυρίως η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ήταν σημαντικό λέγω που βοήθησε στις αποφάσεις αυτές και είμαι ιδιαίτερως ευτυχής που και ε, στην διάσκεψη κορυφής ε, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ε, στην ουσία και ανέθεσαν εις τους αξιωματούχους να βρουν λύσεις μέχρι τον Μάρτιο και το Συμβούλιο Εκοφήν στα τέλη Μαρτίου πήρε την τελική απόφαση και μάλιστα ομόφωνα όπως γνωρίζετε. Ε, και γνωρίζετε βεβαίως ότι για φορολογικά θέματα χρειάζεται ομοφωνία και γι' αυτό η επίτευξη συμφωνιών καμιά φορά είναι εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στον ε, ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Φορολόγησης ε, και το οποίο απέκτησε περαιτέρω ορμή και δύναμη, αν θέλετε, στη διάρκεια της ε, ε, κρίσης, γιατί εκεί φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό να χτυπήσουμε την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή ε, που αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό. Συγκεκριμένα είναι δύο φορές ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πέντε φορές της, του κόστους της κοινή γεωργικής πολιτικής ακριβώς λόγω της κρίσης η οικονομική αλλά και η ηθική και πολιτική σημασία της πάταξης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πρέπει να πω ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων της ε, θητείας μου είδα ότι το θέμα αυτό και στην ε, ατζέντα της Επιτροπής αλλά και στη δικιά μου προσωπική ατζέντα βρισκόταν πάρα πολύ ψηλά. Επομένως, καλή διακυβέρνηση, good governance όσον αφορά την φορολογία. Τον προηγούμενο Ιούνιο, δηλαδή πριν από πολύ μικρόχρονικο μικρό διάστημα το Συμβούλιο Εκοφίνες σε μια ανακοίνωση υπογράμμιζε την σημασία της ε, καλής διακυβέρνησης ε, όσον αφορά την οικονομική πολιτική, όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κυρίως δε και σε διασυνοριακό ε, επίπεδο. Το σημαντικότερο είναι να ε, ενδυναμωθεί η καλή διακυβέρνηση όσον αφορά την φοροδιαφυγή ε, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί χρειάζεται ε, πολιτική βούληση όχι μόνο από τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει πρώτα εμείς να δώσουμε το καλό παράδειγμα γιατί διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να ζητούμε μονάχα από τις τρίτες χώρες καλή διαγωγή ενώ οι δικές μας χώρες έχουν διαγωγή κοσμία Επίσης προωθήθηκαν ε, αυτές ε, οι οδηγίες, όπως ας πούμε για τη διοικητική συνεργασία ή, ε, αυτήν για την αμοιβαία αρρωγή, δηλαδή νομοθετήματα πολύ σημαντικά. Ε, όσον αφορά τώρα τις, ε, την οδηγία για τις ε, εξοικονομήσεις όσον αφορά την φορολογία περιέχουν πολύ σημαντικά στοιχεία για την αποφυγή της στρέβλωσης των αγορών της μείωσης της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής πράγματα επομένως πολύ σημαντικά χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαιτέρως χάρη στην Οικονομική Επιτροπή ε, για την στήριξη της οποίας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου αυτές οι αποφάσεις κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τραπέζι συζήτησης ε, του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ που με τη σειρά του επέτυχε ισορροπημένες πολιτικές αποφάσεις ίδια ε, το φθινόπωρο δηλαδή υπό την Πολωνική Προεδρία. Ε, ε διορθώνω Σουηδική Προεδρία βεβαίως. Ε, θα ήθελα εδώ να αναφερθώ ε, σε δύο συγκεκριμένες ε, τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στις εγγυήσεις των καταθέσεων και στις εγγυήσεις των ασφαλιών και ασφαλιών ζωής κλπ. Γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Μία άλλη σημαντική τροποποίηση είναι η διεύρυνση της νομοθεσίας σε κάποιες σε κάποιους άλλους πόρους καθώς επίσης και σε, κάποιες, σε κάποια άλλα ιδρύματα, funds and foundations. Υπήρξαν και άλλες ε, περαιτέρω θετικές εξελίξεις για τις οποίες θα ήθελα, τις οποίες θα ήθελα να σχολιάσω. Πρώτον, όσον αφορά την εφαρμογή ε, της ε, περικοπής φορολόγησης μέχρι την αυτόματη εφαρμογή, τη, συγγνώμη, την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ήδη από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, ε μία από τις ε, δέκα ε, υπερπόντιες εκτίσεις οι οποίες ανήκουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις κάτω χώρες μεταξύ των οποίων και το νησί του ανθρώπου Island of Man πλέον εμπίπτουν σε ιδιαίτερους κανονισμούς. Επίσης ξεκίνησαν διαβουλεύσεις με τα πέντε με τις πέντε χώρες, Μονακό, Λιχτενστάιν, Σαν Μαρίνο, Ανδόρα ε, και ε, Ελβετική Νομοσπονδία που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Διαβουλεύσεις ξεκίνησαν λοιπόν με τις χώρες αυτές ε, έτσι ώστε να καταλήξουν σε δημιουργείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές αυτών των χωρών με τις αλλαγές στις φορολογικές οδηγίες. Επομένως θα εφαρμόσουν τις τροπολογίες και τις τροποποιήσεις οι χώρες αυτές. Επίσης ξεκίνησαν συζητήσεις με τρία ε, ασιατικά ε, ε, χρηματοοικονομικά κέντρα έτσι ώστε να καλύψουμε και τις κινήσεις προς τις χώρες αυτές Χονγκ Μακάο και Σιγκαπούρη. Αυτά είναι τα τρία χρηματοοικονομικά κέντρα με τα οποία έχουμε ξεκινήσει, με τις οποίες έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις τροποποιήσεις τις οποίες ανέφερα προηγουμένω. Ξέρετε ότι αυτές, ε, ε, οι, αυτά τα κέντρα μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά αρνητικά όσον αφορά οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας για χρηματοοικονομικά ε, ζητήματα και ήδη είναι πολύ θετικό δείγμα το ότι έχουν ξεκινήσει να συζητούν μαζί μας. Επίσης ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με την Νορβηγία η οποία θέλει να προσπογράψει την ε, νέα ε, νομοθεσία. Όλα αυτά που σας αναφέρω είναι θετικές εξελίξεις ευρείας ευρέως γεωγραφικού φάσματος ε, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης έχουμε την οδηγία όπως είπα και προηγουμένως για την αμοιβαία αρρωγή και για την διοικητική συνεργασία. Στις δύο αυτές στα δύο αυτά νομοθετήματα βλέπουμε ότι θα υπάρξει κάλυψη των φορολογουμένων και ε, στις άλλες ε, χώρες. Το απόρριτο εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένες ε, περιπτώσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αποτελέσει πρόσκομα στην ανταλλαγή πληροφοριών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι τροποποιήσεις, οι τροπολογίες τις οποίες αναφέρομαι βρίσκονται ήδη στο τραπέζι του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και ζητώ και από τη δική σας Επιτροπή να στηρίξει τις ε, τροπολογίες αυτές. Ας δούμε τώρα την εξωτερική διάσταση του θέματος. Ένα από τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για την πρόθεση της καλής διακυβέρνησης ε, περί τα φορολογικά είναι οι συμφωνίες ε, με τρίτες χώρες ε, βάση και των προβλεπομένων στο άρθρο 26 ε, των ε, συνθήκων ΩΣΑ και επομένως που οδηγούν στην άρση του τραπεζικού απορρίτου. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις αυτού του είδους με το Λίχτενστάιν και πρέπει να πω ότι το Λίχτενστάιν ήδη μετακινήθηκε από μια θέση απόλυτης μη συνεργασίας σε μια ε, θέση σύμφωνα με την οποία το Λίχτενστάιν είναι πλέον διατεθειμένο να ανταλλάξει ε, πληροφορίες και ενδεχομένως ε, να ε, άρι, το τραπεζικό ε, απόρριτο εάν αυτό αποτελεί ε, εμπόδιο για την περαιτέρω συνεργασία. Επίσης με το Μοναχό, με το Σαν Μαρίνο, με την Ανδόρα και με την Ελβετία ακολουθούμε το ίδιο μοντέλο συνομιλιών και συνεργασίες που είχαμε με το Λίχτενστάιν. Επίσης, σε τέτοιου είδους δεσμεύσεις για ανταλλαγή ε, συνεργασίας ε, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει ε, με διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες. Ακόμα και οικονομικά κίνητρα είναι στη διάθεσή μας έτσι ώστε ορισμένες χώρες της Καραϊβικής και του Ειρηνικού να προχωρήσουν στην προσυπογραφή των αρχών της καλής διακυβέρνησης, ανταλλαγής πληροφοριών κλπ ε, πρόοδος όσον αφορά την, ε, η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των αρχών ανταλλαγών πληροφοριών κτλ. Ε, θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης της φοροδιαφυγής όπου χάνονται δισεκατομμύρια σε επίπεδο ευρωπαϊκό κάθε χρόνο, είναι και αυτό λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο μας είχε απασχολήσει. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο ριζοσπαστικές, πολύ σημαντικές προτάσεις για την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής των ΦΠΑ που, ε, που θα μπορούσε να θεραπεύσει αυτή την απώλεια 67 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μία από αυτές τις προτάσεις, ιδιαίτερα καινοτόμος, επαναστατική θα έλεγα μάλιστα, είναι η πρόταση για την αναστροφή των τελών και η άλλη πρόταση είχε να κάνει με την διακοινωτικη προσφορά, intercommunity supply. Οι δύο αυτές προτάσεις έπρεπε να εξεταστούν από το Συμβούλιο δεν ήμασταν σε θέση εκείνη τη στιγμή να τι εγκρίνουμε τι προτάσει αυτέ στο Συμβούλιο Μομοφωνία. Δεν θελήσαμε όμω να χάσουμε περισσότερο πολύτιμο χρόνο. Επομένω, ε, παραμερίσαμε προσωρινά τις δράσεις αυτές το Δεκέμβριο του 2008 παρουσιάσαμε ένα προσωρινό πρόγραμμα δράσης όπου χρησιμοποιήσαμε μία σειρά από μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και χρησιμοποιούσαν τα κλασικά εθνικά μέτρα εθνικού ελέγχου, εποπτείας, καλύτερες συνεργασίες μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, να γίνει πιο γρήγορη και δώσαμε και ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα, σε δεδομένα ορισμένων βάσεων δεδομένων των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Από τον Δεκέμβριο του 2008 και μετά παρουσιάσαμε το σύνολο των προτάσεων αυτό σε αυτό το προσωρινό σχέδιο δράση με τη μορφή νομοθετική πρόταση στο ΕΚΟΦΗΝ. Επομένω, όλε αυτέ οι προτάσει είναι πλέον επιτάπητο στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και το προτέρημα των προτάσεων αυτών είναι ότι μπορούν τα μέτρα τα οποία περιέχουν να εφαρμοστούν πολύ γρήγορα και δεν παρουσιάζουν κανένα επιπλέον οικονομικό άχθο, ή διοικητικό άχθο για του οικονομικού φορεί. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται νέα ηλεκτρονικά μέσα όπω το e-invoicing, η ηλεκτρονική κοστολόγηση, τιμολόγηση που θα βοηθήσει τη λειτουργία των ε, αρμοδίων φορολογικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης προωθεί το πλήρες σύστημα e-invoice για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε μια εξοικονόμηση 80 εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη. Επίσης, Θέλουμε να έχουμε κοινέ μεθόδου για την καταπολέμηση τη ε, φοροδιαφυγή, για το φόρο προστιθέμενη αξία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναλάβει δράση του κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα μορφή απάτηση. με Την ε, προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε μια νέα πρόταση προκειμένου να χρησιμοποιείται ένα μοντέλο reverse charge, αντιστροφή στελών, αντιστροφής των τελών και να χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πάρα πολλά επίσης είδη, όπως για παράδειγμα τα καλλιντικά ή διάφορα οικιακά είδη ή ε, στους τομείς εκείνους όπου είχε παρατηρηθεί πολύ μεγάλη απάτη στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει υποβληθεί και θα εξεταστεί σύντομα από το Συμβούλιο Κοφίν. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι στα συρτάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΕΚΟΦΗΝ θα αφήσουμε δύο σχέδια προτάσεων τα οποία θα ήθελα εγώ να προωθήσω μια κοινή βάση φορολογική για τις εταιρείε, μια τέτοια πρόταση λοιπόν που έχει ως στόχο να εναρμονίσει όχι την φορολογική βάση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του συστήματος φορολόγησης των εταιριών, αλλά έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα κοινό σύστημα υπολογισμού του εταιρικού φόρου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού της φορολογικής βάσης για τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο οδηγεί σε πάρα πολύ μεγάλες δαπάνες συμμόρφωσης ας συγκρίνουμε την κατάστασή μας με αυτή των ΗΠΑ όπου και οι 50 πολιτείες χρησιμοποιούν μια κοινή μέθοδο υπολογισμού της φορολογική βάσης για τις εταιρείε. Εμείς όπως σας είπα έχουμε 27 διαφορετικά τέτοια συστήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν σε κοινό επίπεδο να έχουμε ένα κοινό σύστημα γιατί αυτό θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητά μας και θα είναι ιδιαίτερα αποφελές για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό εγώ ίδιος θα ήθελα να το προωθήσω τουλάχιστον θα ήθελα να δει το φως ημέρας και ε, μια άλλη πρόταση έχει να κάνει με τη φορολόγηση της ενέργειας. Το ζήτημα αυτό εν μέρη καλύπτεται από το σύστημα εμπορίας των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το σύστημα αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό σίγουρα, αλλά καλύπτει 45% ή έστω και λίγο παραπάνω, γύρω στο 50% των εκπομπών αερίων προκαλούν το θερμοκήπιο. Και το σύστημα αυτό, το εφιστάμενο, δεν καλύπτει προφανώς το υπόλοιπο ίμιση των εκπομπών που δεν καλύπτονται. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε κάποιες μεθόδους οικονομικά αποδοτικές, ένα οικονομικό μέσο προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε τον πολύ αυτοφιλόδοξο στόχο της ε, περιβαλλοντικής ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση δηλαδή κατά 20% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το επίπεδο που είχαμε το 1990 και αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα μέσο λοιπόν το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αγοράς θα ήταν ένα τροποποιημένο σύστημα φορολόγησης ενέργειας. Έχουμε μία ανάλογη οδηγία που έχει να κάνει με το περιεχόμενο της ενέργειας, με το ενεργειακό περιεχόμενο. Εμείς θέλουμε να χωρίσουμε αυτή τη φορολογική βάση σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα θα εξαρτάται από το ενεργειακό περιεχόμενο, ενώ το άλλο τμήμα, όχι απαραίτητα το 50%, θα εξαρτάται από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα προωθηθούν φορολογικά, θα πρημοδοτηθούν φορολογικά οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Αυτή είναι μια δεύτερη πρόταση η οποία θα μπορούσε να προωθηθεί περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι γρήγορα θα περάσει και στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω αυτή τη στιγμή ότι δεν ανλαμβάνω καμία πάγια δέσμευση ε, εξ της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του νέου Επιτρόπου που θα λάβει το χαρτοφυλάκιό μου. Ήθελα απλώς να πω ότι εγώ ίδιος προσωπικά θα ήθελα να προωθηθούν οι δύο αυτές προτάσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Right. Uh, um, σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να βάλω σε τάξη τον κατάλογο των ομιλητών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε δίπλα σας πρέπει να πω κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιλώ ως εισηγήτρια για το ζήτημα της φοροδιαφυγής των τη προστιθέμενης αξίας και όπως και εσείς έτσι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να υιοθετήσουμε μια στάση λίγο πιο φιλόδοξη. Καταλαβαίνουμε όμως ότι πολλές προτάσεις εξαρτώνται τελικά από την ομοφωνία στο Συμβούλιο. Κατάλαβα αυτά που μας είπατε στις προσπάθειες που ε, καταβάλλατε προκειμένου να σταματήσει η φοροδιαφυγή και πώς αυτό επίσης συνδέεται και με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ο κύριος Μάν από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Θέλετε να πάρετε πρώτο το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά που είμαι ο πρώτος που μπορεί να θέσει ερωτήσεις. Κύριε Κόβατσα, έχουμε πολλά σύμφωνοι εγώ τώρα στο θέμα των, του κλεισίματος ή της συρρήκνωσης των ε, οάσεων των φορολογικών. Το έχουμε εγγράψει εδώ και χρόνια στην ημερησία διάταξη και υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Όποτε γίνεται κάτι παραγωγικό δίνεται η απάντηση δεν επαρκεί αυτό. Οι άλλοι λένε τι ωφελεί τώρα στο Λίχτερστάιν να έχουμε κάποιες αλλαγές στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία και αλλού. Και να υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογών όταν σε άλλα μέρη του κόσμου αυτά δεν λειτουργούν, στη Σιγκαπούρη για παράδειγμα. Ε, τότε θα τοποθετήσουμε, λέει, και θα επενδύσουμε αυτά τα χρήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε να καλύψουμε και αυτά. Είπατε, τα πρώτα βήματα γίνονται. Πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση. Πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση να καταφέρουμε να συμμετάσχουν σε αυτά τα μέτρα και άλλες χώρες. Να έχουν φορολογική συνεργασία οι αρχές δίωξη τη αφοροαπάτης από αρχέ όπου δεν είχαν συνεργασία στο παρελθόν και να υπάρχει μια στρατηγική αποτροπή... Ε, ή αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή είναι κάτι που θα έπρεπε να προχωρήσει και να μάθουν από την Ευρώπη. Και το θέμα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Είπατε στο τέλο τη εντολή σα φτάσατε. Τώρα δεν ξέρουμε το τι θα γίνει συνέχεια. Μπορεί να μάθει το Συμβούλιο Υπουργών ΕΚΟΦΗΝ κάτι. Μπορούν να το μάθουν όχι επειδή έχουμε μια κρίση στην οποία πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά θέλουμε να μάθουμε ένα από τον άλλο, διότι είναι θέμα ορθολογικό είναι θέμα λογικής να έχουμε κοινού κανόνες και να προσπαθήσουμε θελοντικά ο ένας να ανταποκριθεί στα αιτήματα του άλλου. Υπάρχει αυτή η βούληση να, για μάθηση και να μάθουν τελευταία ερώτηση για το ΦΠΑ και τις ε, αλλαγές. Το είδαμε στη χώρα μου οι μικρές επιχειρήσεις έχουν τεράστια ε, δυνατότητα και ευκαιρία να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εντάξει, συμφωνώ, ήταν επιτυχές το μέτρο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παντού, λένε άλλοι, μειωμένα ποσοστά, να έχουμε μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ μπορεί κανείς να μάθει, ποια είναι η σωστή οδός να μάθει κανείς. Να μάθουμε, όχι επειδή είναι μια κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να μάθουμε με τους άλλους για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αποτελεσματικά όλοι. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτον όσον αφορά τις φορολογικές οάσεις, να πω ότι καθότι γνωρίζω σχετικά οι φοροάσεις σε κάποιες χώρες. Στη χώρα που γνωρίζω εγώ καλύτερα για παράδειγμα υπάρχουν κάποιες απόψεις που λένε ότι οι φοροάσεις είναι μια περιοχή όπου ο αντίπαλος μου, ο πολιτικός μου αντίπαλος έχει επενδύσει εκεί. Υπάρχουν όμως και αντικειμενικά κριτήρια, πολύ πιο αντικειμενικά από αυτή την αξιολόγηση. Πρώτον, φοροάσεις είναι ένας τόπος όπου η φορολογία είναι υπερβολικά περίπλοκη και σίγουρα όχι ε, διαφανής. Δεύτερον, φοροάσεις με διακριτική ευχέρεια επιβάλλεται φορολογία, χαμηλή φορολογία, χαμηλότερη φορολογία για τους επενδυτές από ό,τι για τους Ιθαγενείς για να συλλέξουν κεφάλαια. Και τρίτον, οι φοροάσεις είναι ένα μέρος όπου ποτέ δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες ε, όσον αφορά θέματα φορολογουμένου και αναφέρονται στο τραπεζικό απόρριτο πάντα όταν ζητούνται τέτοια στοιχεία. Αυτό είναι το επιχείρημά τους γιατί δεν μπορούν να δώσουν τέτοιες πληροφορίες. Αυτά είναι τρία λοιπόν αντικειμενικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν τις φοροάσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι περίεργο να πει κανεί ε, ότι επειδή έχει τεράστια αρνητική επίπτωση η κρίση στις οικονομίες μας γίνεται αυτό. Αλλά κάποιο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι η πολιτική βούληση που απέρευσε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα, να αντιμετωπιστούν και επιληθούν, να μειωθεί η φοροαπάτη, η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή και να καταφέρουμε να πετύχουμε η καταπολέμηση των φοροάσεων να είναι πιο ε, δραστήρια, ε, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και να προχωρήσει ως θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ σημαντικό ρόλο να ε, διαδραματίσει σε σχέση με τέτοιες προτάσεις και πρωτοβουλίες. Δεν θα είμαστε επιτυχείς αν δεν είχαμε υποστηριχθεί από τα κράτη-μέλη σίγουρα και επίσης από χώρες όπως από τις χώρες της Λέσχης των 20 της ε, Group 20. Θυμάμαι όταν προπαρασκευαζόταν τον Απρίλιο αυτή η Σύνοδος Κορυφής της Λέσχης των 20 και κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες ήταν σαφές ότι η Λέσχη των 20 θα ήταν πρόθυμη να επιβάλλει κυρώσεις κατά των μη συνεργάσιμων αρχών. Σε λίγες εβδομάδες τουλάχιστον 40 διαφορετικές ε, αρχές που είχαν εγγραφεί στον ε, φεό κατάλογο του ΩΣΑ έστειλαν μήνυμα και ανέφεραν ότι έχουν υιοθετήσει μια νέα θέση και θα ήταν πρόθυμες να συνεργαστούν σύμφωνα με το άρθρο 26 της ε, πρότυπης σύμβασης ΩΣΑ. Πολλές ε, νήσεις στον Ατλαντικό ωκεανό, στον Ειρηνικό ωκεανό, στην Καραϊβική και υπηρετικές ε, χώρες επίσης. Και σίγουρα αυτό ήταν ένα πολύ καλό θετικό μήνυμα Ακόμα και μετά τη Σύνοδο του Λονδίνου πήγα στο Παρίσι για να έχω επαφές και συζητήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων έφτασε ένα μήνυμα ότι οι τελευταίες χώρες του Μαυροπίνακα, νομίζω Παναμάς, Κωνσταντίνα, Φιλιππίνες και η Μαλαισία ήταν αυτές οι τέσσερις χώρες. Ανήγγυλαν λοιπόν αυτές οι τέσσερις χώρες ότι θα ήταν πρόθυμες εφ' εξής να συνεργαστούν. Δεν υπάρχει λοιπόν πια μαύρο Δεν υπάρχει ούτε καν φεός πίνακας, γκρίζος πίνακας. Υπάρχει ένας αριθμός χωρών που ανέφεραν ότι δεσμεύονται να συμμορφωθούν με, αυτή, με αυτές τις αρχές. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές από αυτές τις χώρες λένε ότι είναι πρόθυμες να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια του 2002-2003 και δεν συμμορφώθηκαν, δεν υλοποίησαν αυτή την υπόσχεσή τους, δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους. Συμφωνούμε λοιπόν με τον ΟΣΑ και με τη γραμματεία του ΟΣΑ ότι η Γραμματεία του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επισκοπήσουν, να επιτηρήσουν σαφώ την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων από αυτέ τι χώρε. Και με ικανοποίηση σημείωσα ότι κατά τι τελευταίε συνεδριάσεις της Λέσχη των 20 στη Σύνοδο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αυτό που έκαναν ήταν και πάλι επιβεβαίωσαν την δέσμευση που ανέλαβαν, είχαν αναλάβει, ώστε την επόμενη, μέχρι την επόμενη άνοιξη να ε, ληφθούν μέτρα κατά όλων εκείνων που δεν ε, συμμορφώνονται με αυτές τις διατάξεις. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο. Αναφέρατε εξειδικευμένα συγκεκριμένα την Σιγκαπούρη. Να απαντήσω με ένα άλλο παράδειγμα, το Χονγκ Κονγκ που το γνωρίζω καλύτερα. Είχα και προσωπικά διαπραγματευτεί, αλλά νομίζω εντάσσονται στην ίδια κατηγορία. Όταν πήγα για πρώτη φορά με του συναδέλφου μου στο Χονγκ Κονγκ, τι συνέβη. Ο Υπουργό Οικονομικών του Χονγκ Κονγκ επιχειρηματολογούσε και έλεγε δεν μπορούν λέει, να ανταλλάξουν τέτοιου είδου πληροφορίε πρώτα και κύρια επειδή δεν φορολογούν λέει τις αποταμιεύσεις είτε αποταμιεύσεις ε, ε, κατοίκων, μονίμων κατοίκων ή και μη κατοίκων και σαν συνέπεια αυτού δεν συλλέγουν πληροφοριακά στοιχεία και καθώς δεν συλλέγουν δεν έχουν τίποτα να ανταλλάξουν ακόμα και αν είχαν λέει τέτοια στοιχεία η νομοθεσία του Hong Kong δεν θα επέτρεπε να ανταλλάξουν αυτά τα στοιχεία και δεν υπάρχει λοιπόν αντικείμενο συζήτησης είχαν πει και το θέμα έλυγε. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά τι έγινε. Ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών προσήλθε στις Βρυξέλλες, στο γραφείο μου και εξέφρασε ο ίδιος τη βούληση πλήρως να συνεργαστεί το Χονγκ Κονγκ και τη συμμετοχή του, συμμετοχή του ως Χονγκ Κονγκ στις ρυθμίσεις για φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι' αυτό. Τώρα, σε σχέση με το άλλο θέμα για τον μη εξαντλητικό πίνακα που ήταν συμβιβασμός και έπρεπε να εργαστώ εργοδός ε, με μεγάλο κόπο εργάστηκα για να τα καταφέρω να υπάρξουν συμφωνίες με εκείνα τα κράτη-μέλη που έλεγαν ναι υποστηρίζουμε αυτή την ιδέα αν όμως επιτευχθεί αυτό ή το άλλο ως ε, ε, ανταπόκριση και αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ φυσικά να βλάπτει τα συμφέροντα άλλων κρατών μελών. Τώρα, το σημείο κλειδί ποιο είναι. Είναι μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ δεν είναι υποχρεωτικά. Είναι μια εναλλακτική λύση. Εθελοντικά μπορούν να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη. Ε, σε σχέση με τις υπηρεσίες και κάποια αγαθά για μειωμένα τέτοια ποσοστά ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την επίκαιρη, επικαιροποιημένη κατάστασή τους ε, τα κράτη-μέλη μπορούν ή μπορούν να εφαρμόσουν αυτόν τον κατάλογο με περιορισμένο ε, ποσοστό ΦΠΑ ή και μπορούν να μην τον εφαρμόσουν. Ευχαριστώ Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Και τώρα, τώρα σε σχέση με τις άλλες ε, παρατηρήσεις έχουμε έναν ολόκληρο κατάλογο 15 ατόμων που περιμένουν να παρέμβουν. Ο πρώτος για την ομάδα SD είναι ο κύριος Ντομινίτσι νομίζω. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Κόβατς. Είπατε, συνοψίζοντας ε, ή εν συμπεράσματι μάλλον, είναι ότι δεν ξέρετε τι θα γίνει στο μέλλον. Όμως ε, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσατε ε, και τα οποία απαιτούν και προϋποθέτουν οπωσδήποτε κάποιες, κά, κάποιες οδηγίες που θα ακολουθήσει και η επόμενη ε, Επιτροπή, κυρίως οτιδήποτε σχετίζεται με την φορολογική good governance. Εάν εμείς αναφερόμαστε στην καλή διακυβέρνηση ε, με πλαίσια διαφάνειας, ε, ανταλλαγής πληροφοριών κτλ, οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί σαν καλή δουλειά και για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία, αναφέρομαι ιδιαίτερως στο πλήρες ξεπέρασμα μετά από πρόταση και δική Τη ε, την, ε, της άρσης του τραπεζικού απορρίτου για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για, τις, για τους μη αυτόχθονες, μη γηγενείς σε άλλες χώρες. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα της ε, αμοιβαίας ε, αρρωγής, ε, της δυνατότητα συνεργασίας, διοικητής συνεργασίας με αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς επίσης και την συνεργασία όσον αφορά την αποταμίευση και όσον αφορά και τις ειδικέ μορφές επενδύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά τα θέματα να μιλάει με μία φωνή. Είναι θετικό λοιπόν που ε, ότι πολλές χώρες ε, έχουν προσυπογράψει τις αρχές ε, του ΩΣΑ. Αλλά είπατε κι εσείς ο ίδιος ότι αυτή η προσυπογραφή πολύ συχνά δεν ακολουθείται από ενσωμάτωση των αρχών αυτών στην νομοθεσία των εν λόγω κρατών και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σε περίπτωση ενσωμάτωσης, πολύ συχνά ε, τα, ε, οι εφαρμοστικοί κανόνες δεν είναι τέτοιοι που να επιτρέπουν εύκολη και άμεση εφαρμογή. Επίσης πιστεύω ότι η εποπτεία, το monitoring και ο έλεγχος θα πρέπει να είναι ε, συνεχής και επομένως πιστεύω ότι οι αρχές σε καλής διακυβέρνησης, good governance, θα πρέπει να αποτελεί συγκεκριμένο κεφάλαιο το οποίο θα αναφέρεται σε οποιαδήποτε διμερή ή πολυμερή συμφωνία με τρίτες χώρες, κυρίως δε με αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί πιστεύω ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι η προώθηση τυποποιημένων συστημάτων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτά λοιπόν είναι ορισμένα πολύ θετικά και σημαντικά στοιχεία. Εγώ σας ρωτώ επίσης, ε, επί δύο συγκεκριμένων ζητημάτων, ποια είναι η θέση σας. Τούτη τη στιγμή γίνεται λόγος αλλά και στην πράξη εφαρμόζονται, ε, ακούγονται κάποιες ε, κινήσεις για την αμνηστία, αν θέλετε, για τον επαναπατρισμό ε, κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Αυτό που ονομάζουμε φορολογική ασπίδα. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Δεν πιστεύετε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει συντονισμός όσον αφορά τα βασικά κριτήρια που θα ισχύσουν για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ποια είναι η άποψή ε, σχετικά με το να υπάρξει ένα γενικότερο πλαίσιο όσον αφορά την φορολόγηση των ε, χρηματοοικονομικών κινήσεων και συναλλαγών. Απάντηση. Ναι, είναι γεγονός ότι στο τέλος της εισήγησής μου ε, αναφέρθηκα στο CCCTB Ε, είναι γεγονός ότι ε, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ τα αφήνω στο ψυγείο. Όμως θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως η καλή διακυβέρνηση, η good governance όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα δεν είναι καθόλου στο ψυγείο, δεν είναι καθόλου στα χρονοτούλαπα. Είναι ε, πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων και επομένω ε, θα συνεχιστεί η συζήτηση. Απλώς εγώ δεν μπορώ να αναλάβω καμία δέσμευση για την επόμενη επιτροπή, για το επόμενο ε, σχήμα όσον αφορά το CCTB και την συγκεκριμένη μορφή που θα πάρει. και από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι αυτού του είδους ε, η ε, καλή συνεργασία και ε, θα πρέπει πρώτα να γίνει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την απαιτήσουμε και από το, από το εξωτερικό της. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά. Ε, όμως πρέπει να σας πω επίσης ότι και η γραμματεία του ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευτεί και μαζί και το, το G20 να έχουν κάποια κοινή πορεία όσον αφορά την ε, φορολογία και όσον αφορά και την ανταλλαγή, ε, την ανταλλαγή πληροφοριών και το τραπεζικό απόρριτο και αυτό είναι ε, πολλά υποσχόμενο για το μέλλον. Αναφέρετε το γεγονός ότι κατά την άποψή σα θα πρέπει να αναφέρετε μια, σε μια παράγραφο η καλή ε, διακυβέρνηση σε οποιασδήποτε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες. Μα ακριβώς αυτή είναι η πολυμερεις συμφωνιες μα ακριβώ αυτη ειναι η προθεση μας. Ακριβώς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία κάνουν, ε, οποιαδήποτε διμερή συμφωνία κάνουν οι χώρε μέλη να περιλαμβάνουν και μια τέτοιου είδου παράγραφο. Νομίζω ότι απήντησα στις ερωτήσεις σας. Α, όχι, είπατε και για τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτή η ιδέα έρχεται και φεύγει, ξαναεμφανίζεται στο προσκήνιο. Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών, και τον ρόλο που έπαιξαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αυτήν την κρίση, νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό που επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη. Ήδη πριν από μερικά χρόνια ξανά ήταν στην ατζέντα μας. Ε, ε, δηλαδή αναφερόμαστε σε ένα είδος συνέχεια της, συνέχεια της Tobin ε, Tax, λαμβάνοντας υπόψη και κάποια νέα ε, στοιχεία, νέα δεδομένα. Δεν υπάρχει ακόμα νομοθετική μορφή. θέλουμε όμως μια γενική αρχή η οποία να ακολουθεί ακριβώς αυτά τα δεδομένα. σίγουρα θα μπορούσε να να δώσει κάποια επιπλέον έσοδα στον κοινοτικό ε, προϋπολογισμό. Όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, για όλα τα φορολογικά χρειάζεται ομοφωνία ε, και διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το κατά πόσον μια τέτοιου είδους απόφαση θα ετύχανε ομοφωνίας. Ε, με ναι. ρωτήσατε κάτι άλλο? Α, ναι, ναι, αμνηστία, φορολογική αμνηστία. Όχι, δεν είναι, αυτό δεν είναι ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη μπορώ να σας την πω. αλλά μονάχα σαν άτομο και, σαν, ε, και όχι σαν επίτροπος. Εγώ, λοιπόν, συμμερίζομαι τις απόψεις αυτών και δεν αναφέρομαι στην Ιταλία τώρα, αναφέρομαι ε, σε όλες τις ε, χώρες. Ε, υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι αυτού του είδους η αμνηστία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια, ένα δεοντολογικό κενό ή κάποια ηθική αμφιβολία, αν θέλετε, στο μεγάλο σώμα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Κουίντς από την ομάδα Άλντι. Ναι κύριε Πίτροπε, από την εισαγωγή σας κατανόησα ότι δεν υπολογίζετε να ανήκετε πάλι στη νέα Επιτροπή. Ίσως είναι αυτή λοιπόν η τελευταία μας συνάντηση εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που καταβάλατε και που καταδείξατε με σαφήνεια ποιοι είναι οι στόχοι σας. Τώρα, κατά πόσον αυτή η προσπάθεια θα στεφθεί, στέφτε με επιτυχία, θα το δείξουν τα επόμενα χρόνια στο μέλλον. Πολλά έγιναν προσπάθεια να επιτευχθούν, αλλά καταδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολο στον τομέα της φορολογίας να σημειώσει κανείς πρόοδο, πραγματική πρόοδο. Δύο-τρία σχόλια πρώτα και κάποιες ερωτήσεις μετά. Μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ. Εγώ θεωρώ ότι δεν υλοποίησε αυτό, πιστεύω, αυτά τα οποία ελπίζαμε. Εγώ ίδιος στην Γαλλία πρόσφατα είδα προσωπικά πώς οι εστιατόρες αυτή τη μείωση την χρησιμοποίησαν για μείωση τιμών. Πολύ περιθωριακό ήταν αυτό. Ίσως σε κάποια γεύματα, σε κάποια ε, πιάτα υπήρχε κάποια τέτοια μικρή μείωση. Πόσο πραγματικά όμως ε, πάει στην ίδια τσέπη και πόσο υποφελούνται οι καταναλωτές, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τολμώ να απαντήσω. Μάλλον 50-50, ας μην υπερεκτιμούμε όμως το αποτέλεσμα του μειωμένου ποσοστού ΦΠΑ. Τώρα το δεύτερο σημείο αφορά τις απάτες, φοροαπάτες πρέπει να πω εδώ ακόμα δεν μπορώ τα δύο αυτά να τα συνδυάσω μεταξύ του ποσού που αναφέρατε συμπεριλαμβανομένης της απάτης ΦΠΑ 250 δις ευρώ ετήσια είπατε και του ποσού εκείνου που με την ε, υποχρέωση ανακοινώσεων ή ανταλλαγής ε, στοιχείων κατά των ε, φοροάσεων τι μπορεί να επιτευχθεί. Αν δούμε αυτά τα μεγέθη τότε είναι περιθωριακά από τα τεράστια ποσά και κονδύλια που διακινούνται. Θα έπρεπε μεγαλύτερο ποσοστό. Ε, βλέπουμε ότι 90% παρακάμπτει καν τη φορολογία και δεν φορολογείται είτε είναι Λίχτενστάιν, Ελβετία, Βέλγιο, οπουδήποτε αν πηγαίνουν κάπου αλλού και δεν φορολογούνται. Και είναι ευχάριστο το ότι όλοι λένε ότι είναι πρόθυμοι πραγματικά να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή αυτών των στοιχείων για την καταπολέμηση της φοροαπάτης. Παρόλα αυτά όμως τα έσοδα βρίσκονται πολύ πιο πίσω από αυτά που θα έπρεπε να ήταν. Αλλά τέλος πάντων εσείς δεν μπορείτε να τα αλλάξετε αυτά. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είδαμε ότι στην εποπτεία είχαμε regulatory arbitrage, δηλαδή οι συμμετέχοντες στην αγορά γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι θα έπρεπε να κάνουν ώστε να υποφεληθούν από διαφορές σε σχέση με την εποπτεία. Και το ίδιο ισχύει και με τη φορολόγηση. Όσοι εμπλέκονται στην αγορά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να υποφελούνται από διαφορετικές διατάξεις για τη φορολογία. Πρώτον, πώς φορολογούνται διαφορετικά και πώς μπορούν να ξεφύγουν από τη φορολογία αυτή θα έπρεπε να είχαμε καταλάβει ότι παράλληλα με το regulatory arbitrage το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με νέε δομέ στην εποπτεία και στην επιτήρηση ώστε στην Ευρώπη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο αλλά και στου φόρου να κάνουμε κάτι παρόμοιο, στη φορολογία. Κατά του tax arbitrage πρέπει να γίνει κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ποσοστά φορολογία θα είναι εξομοιωμένα και θα είναι τα ίδια, αλλά τουλάχιστον από πλευρά δομή θα πρέπει να είναι καλύτερα συγκρίσιμα αυτά τα στοιχεία για τη φορολογία από ό,τι σήμερα. Και διαρωτώ με δεν θα έπρεπε να προβληματιστούμε και να δούμε και εγώ είμαι υπέρ φιλελεύθερα υπέρ του φορολογικού ανταγωνισμού. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά το ΦΠΑ δεν θα έπρεπε να υπάρξει σαφέστερα εναρμονισμός από ότι αυτός που υπάρχει σήμερα. Τώρα, μεταξύ 15 και 20% λένε. Είναι μεγάλη διαφορά αυτή η ψαλίδα. Θα ήθελα να φτάσουμε πιο κοντά στα όρια. Διότι ένα είναι βέβαιο, με τον βαθμό υπερχρέωση στα κράτη-μέλη, ενδιαφέρον θα ήταν να είχαμε ένα ενιαίο ποσοστό ΦΠΑ. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη τώρα ως μικροεπενδυτής διαπιστώνω το εξής. Αν έχω μια μετοχή της Nokia στη Φινλανδία και μου δίνει μέρισμα, μου καταβάλει μέρισμα η Nokia και έτσι παίρνει ε, κάποια ποσά η Φινλανδία. Μπορώ να τα υπολογίσω αυτά ή όταν υποβάλω τη φορολογική μου δήλωση να μου επιστραφούν. Αν έχω μια μετοχή της UBS στην Ελβετία, το ίδιο. Τώρα, τα φορολογικά ποσοστά διαφέρουν στο ύψο του, αλλά το πολύ χειρότερο είναι, αυτό δεν είναι τίποτα τρομερό, διότι μου επιστρέφουν μέρο τη φορολογία. αλλά η διαδικασία πώ μου επιστρέφονται αυτά τα ποσοστά φορολόγηση είναι τελείω διαφορετικέ οι διαδικασίε από τη μια χώρα στην άλλη. Και είναι τόσο μεγάλη η γραφειοκρατική ε, επιβάρυνση που στο τέλο λέει κανεί, «Ε, πάει στα τσακίδια να απεμπολίσω αυτά τα 10-15% που θα μου επιστραφούν μια και είναι τόσο περίπλοκες και ε, παχθείς οι διαδικασίες. Εδώ θα έπρεπε να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι ώστε να διασφαλίσει ότι πραγματικά για τους μικροεπενδυτές θα είναι λειτουργούσα η κατάσταση και όχι δυσλειτουργική. Yes, I ε, Μάλιστα. Συμφωνώ με την άποψή σας ότι στα πλαίσια της φορολογίας είναι πολύ δύσκολο να καινοτομήσει κανείς. Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λένε, λέτε, το είδα και εγώ κατά τη διάρκεια της πεντετούς ε, θητείας μου. Ωστόσο, θεωρώ ότι πετύχαμε κάτι το οποίο ελάχιστη περίμενα ότι το καταφέρναμε. Όσον αφορά τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ, συμφωνώ μαζί σας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα μειωμένα ποσοστά δεν μεταφέρονται στη συνέχεια στον καταναλωτή Ακόμα και οι αυξήσει όμως στη φορολογία δεν μεταφέρονται εξαιτία του ανταγωνισμού. Η εφαρμογή όμω των μειωμένων ποσοστών δεν ήταν μια εναλλακτική λύση. Αυτό ήταν το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποίησα όταν χρειάστηκε να πείσω κάποια κράτη-μέλη όπως η Γερμανία, η Ιδανία και κάποιες άλλες χώρες οι οποίε δεν θέλουν καμία επέκταση του καταλόγου για τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο εγώ συμμετείχα τόσο πολύ και ασκούσα πίεση ήταν γιατί ήθελα να δώσω τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερη περιθώρια ευελιξίας μέσω της επιλογής που θα είχαν. Δεν νομίζω όμως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο στο μέλλον, γιατί ε, στο εκοφήν του Μαρτίου η γενικότερη στάση των κρατών μελών ήταν ενάντια στην πρόταση αυτή των μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ. Και στο υπόλοιπο της θητείας μου δεν έχω σαφώς το χρόνο για να υποβάλω κάποια νέα πρόταση. Μία σημαντική πάντως πρόταση η οποία δεν ευωδόθηκε ήταν η εφαρμογή των μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ στα πράσινα προϊόντα, πρόταση των Βρετανών και των Γάλλων η οποία όμως τελικά δεν στέφθηκε με επιτυχία στο τελευταίο κοφήν του Μαρτίου. Δεν παρουσιάστηκε καν, δεν έφτασε καν στο σημείο της παρουσίασης. Όσον αφορά τώρα την φοροαπάτη, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ βήμα προς βήμα και νομίζω ότι ήδη έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε μια σημαντική πρόοδο. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν φτάσαμε ε, τα μηδενικά ποσοστά φορολογικής απάτης, παρόλα αυτά η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό το οποίο μας βοήθησε είναι ότι η ίδια η κρίση βέβαια, η χρηματοοικονομική κρίση, καθώς επίσης ε, και οι νέες πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση. Όσον αφορά τώρα την ε, εναρμόνιση του φόρου προστιθέμενης αξίας, ένας ενιαίο ποσοστό. Πρέπει να σας πω προς αυτό ότι κάναμε μία μελέτη, έκανε μία μελέτη μάλλον μία ανεξάρτητη, ένα εξάρτητος οικονομικός φορέας, ο οποίος μελέτησε το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης ενός ενιαίου ποσοστού και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από οικονομικής πλευράς η πιο λογική λύση θα ήταν υπάρχει ένα και μοναδικό ποσοστό σε κάθε χώρα. Όχι το ίδιο ποσοστό φορολογικό ΦΠΑ για όλες τις χώρες, αλλά το ίδιο στο στερικό κάθε χώρας. Για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους όπως η απασχόληση, όπως ο πολιτισμός, όπως τα audiobooks για παράδειγμα. Συμπεριλήφθηκαν και κάποια προϊόντα από τους τομείς αυτούς ή υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγειονομική περίθαλψη ή ακόμα και πολιτική περιβάλλοντος. Προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς αυτούς θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από τη χρησιμοποίηση ενός ενιαίου α, ποσοστού. Επίσης η εταιρεία αυτή, ο οικονομικός αυτός φορέας μας είπε ότι ε, δεν θα ήταν ε, σωστό μόνο από οικονομικής πλευράς να υπάρχει ένας ενιαίος συντελεστής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ένα ελάχιστο ποσοστό, ένα ελάχιστο τελεστή τη τάξη του 5%. Στον αφορά το παράδειγμα με την όκια το οποίο μας παραθέσατε, θα το εξετάσουμε περισσότερο και θα σας δώσουμε μια απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Από την ομάδα των συντηρητικών, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Uh, Εγώ είμαι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου ήδη στην αρχή αρχή να σας ευχαριστήσω για αυτή την πενταετία που συνεργαστήκαμε τόσο, συνεργαστήκατε τόσο στενά με την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Πιστεύω ότι πολύ σωστά δράσατε όσον αφορά τον τομέα της φορολογίας. Γνωρίζω και έχω συνειδητοποιήσει, Πρόεδρε, ότι υπάρχει μεγάλος κατάλογος αγορητών. Θα είμαι λοιπόν όσο δυνατόν συντομότερος. Η ερώτησή μου είναι λοιπόν, είναι εύκολη θα έλεγα εύληπτη για την Common Consolidated Tax Base, το CCTB. Συμμερίζομαι την ίδια άποψη για τον φοροανταγωνισμό όπως ο προλαλή σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω και όχι υπό τεχνικής, από τεχνικής πλευράς δεν θέλω να κάνουμε λόγο για τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες ε, των, του, του Τα καλά μαντάτα είναι ότι αυτή η πρόταση απέμεινε στο τραπέζι σας, στο γραφείο σας και θα συζητηθεί στη συνέχεια, ελπίζω ότι θα γίνει αυτό, στο απότερο μέλλον, έστω. Αλλά τι πιστεύετε εσείς προσωπικά, ποια είναι η ατμόσφαιρα, το κλίμα στο ΕΚΟΦΗΝ ποια είναι η διάθεση, ας το πούμε έτσι, η βούληση των κρατών μελών για, επ' αυτής της προτάσεως που είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντική για το μέλλον. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ εκ προημίου για την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Το 2006, κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, τον Αυστριακό Υπουργό Οικονομικών. Είχα ζητήσει να το εγγράψει στην ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη ενός άτυπου συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και να το εγγράψει ακόμα πιο άτυπα στην, ε, στο μενού του ε, γεύματός μας. Ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητικό να ακούσει κανείς τις απόψεις ε, των 27 εκπροσώπων των κρατών μελών Υπουργών Οικονομικών. Τότε ήταν 25 μόνο τα κράτη-μέλη, πριν από την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας <clears throat> αλλά ήταν παρόντες ως παρατητές και ξέφρασαν απόψεις λοιπόν. Παρόλα αυτά, αν θυμάμαι σωστά, 12 κράτη-μέλη ήταν έντονα υπέρ και μάλιστα παρότριναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απίθυναν έκκληση να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο μακριά και όσο το δυνατόν ταχύτερα. Δέκα περίπου κράτη-μέλη ήταν προσεκτικά, επιφυλακτικά, υποστηρικτικά δεν είχε υποβληθεί απλά, ε, δεν είχε υποβληθεί κάποια νομική πρόταση με νομική βάση, μια πρόταση γενικά είχε τεθεί επί τραπέζης. Έξι όμως όμως μέλη είχαν εκφράσει ανησυχίες Κάποιες χώρες έλεγαν ότι θα ήταν παραβίαση όσον αφορά τα κυριαρχικά φορολογικά δικαιώματα κρατών μελών. Η απάντησή μου ήταν δεν θα υπήρχε καμία τέτοια παραβίαση κυριαρχικών φορολογικών δικαιωμάτων κράτους μέλους. Διότι το να καθορίσουν τα ποσοστά ΦΠΑ θα παρέμενε αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα μπορούσαν να διατηρήσουν λοιπόν τα θέματα φορολογικής κυριαρχίας τους, κυριαρχικά δικαιώματα. Κάποιες χώρες είπαν ότι θα ακολουθούσε σύντομα ο εναρμονισμός ποσοστών φορολόγησης και εγώ ορκίστηκα ότι δεν, δεν ήταν καν στην πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Επιτρόπου κάτι τέτοιο να τερματιστεί ο φοροανταγωνισμός διότι ο φοροανταγωνισμός έχει ωφέλη σίγουρα είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, το τρίτο επιχείρημα, και αυτό ήταν το πιο ορθολογικού χαρακτήρα επιχείρημα, ήταν εκείνο που προήλθε από χώρες όπως για παράδειγμα της ε, Βαλτικής ή της Σλοβακία, τη Σλοβακία που έχουν ένα ενιαίο ποσοστό φορολόγησης είχαν εκφράσει την ανησυχία τους ότι μια νέα εναρμονισμένη φορολογική βάση θα ήταν λιγότερο ευρεία από ότι η φορολογική βάση που χρησιμοποιούσαν, που ήταν ευρύτερη. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον ε, Υπουργό Οικονομικών της Σλοβακίας είχε εκφραστεί του πατέρα του ενιαίου συστήματος φορολόγησης στη Σλοβακία. Τώρα, η πρότασή μου ήταν υπέρ της συγκεκριμένης αυτής πρότασης διότι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να υπάρχει ευρύτατη, απλούστατη, όσο το δυνατόν ε, φορολογική βάση ή δυνατόν χωρίς καμιά εξαίρεση ή με ελάχιστες εξαιρέσεις και είπαν τότε κάποιοι ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα μπορούσε η με ελάχιστε εξαιρέσει. Και είπαν τότε κάποιοι ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο θα μπορούσε η Σλοβακία να επανεξετάσει τη θέση τη ε, και ίσω να την αναθεωρήσει. Αυτά έμαθα τότε και ήταν πολύ επικοδομητική διδα... δι... από πλευρά ε, διδαχή ε, επικοδομητικό το εγχείρημα. Είχα την ελπίδα ότι κάποτε θα μπορούσαμε να έχουμε ομοφωνία, να πετύχουμε μια τέτοια συμφωνία για διευρυμένη συμμετοχή και συνεργασία 18-20 21, 22 ίσως χωρών. Αλλά αυτό είναι φυσικά, θα είναι η αρμοδιότητα, η ευθύνη του επόμενου επιτρόπου στην επόμενη νέα ε, επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο πρώτος των Πρασίνων. Παρακαλώ εσείς. First of all... Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Επίτροπε. Μεγάλη εκτίμηση υπάρχει στην ομάδα μας για την εργασία σας, το έργο σας, παρότι ακόμα μπορεί να υπάρχουν κάποιες φιλοσοφικού χαρακτήρα διαφορές όσον αφορά τον ρόλο του φοροανταγωνισμού. Εκτιμούμε όμως ιδιαίτερα το έργο που επιτελέσατε. Και για το γεγονός επίσης ότι οι επιζήμιες μορφές ε, φοροανταγωνισμού εξακολουθούν να είναι τόσο σημαντικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συμβαίνει όχι επειδή εσείς είχατε ελλείψεις ε, ή δεν είσαστε πλήρης ε, στην δράση σας, αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης από άλλους οφείλεται σε άλλους λοιπόν. Πιστεύουμε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής θα είναι όλο και περισσότερη, όλο και σημαντικότερη τα επόμενα χρόνια διότι οι απώλειες από πλευράς εσόδων στον προϋπολογισμό και το χαμηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας όσον αφορά τα φοροέσοδα θα είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή και είναι σίγουρο ότι οπωσδήποτε αυτή η κατάσταση θα αποτελέσει έναυσμα για να σημειωθεί επιτέλους πρόοδος. Τρεις σύντομες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μετά από αίτημα δεν επαρκεί. Και γι' αυτό έχουμε την οδηγία περί αποταμίευσεων, την αρχή της αυτόματης ανταλλαγής ε, στοιχείων. Και αυτό θα πρέπει να επεκταθεί, να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Ερώτηση. Υπήρξαν κάποτε διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και τη συμμόρφωση με αυτή την αρχή και με ποια επιτυχία έγινε αυτό. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπήρξαν άτυπα ή επίσημα επαφές για τέτοια αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων σε θέματα φορολογίας. Δεύτερον, έχουμε ένα δεοντολογικό κώδικα για τη, τη φορολογία επιχειρήσεων. Ακόμα και αν το CCTB, το Common Consolidated Tax Base, δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα, έχουμε τον δεοντολογικό κώδικα. Με αυτόν έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Πολλά όμω κράτη-μέλη βρήκαν νέους τρόπους να παρακάμπτουν, α το πω έτσι, τον δεοντολογικό κώδικα και με μεγάλες απώλειες επιπλέον για πολλά κράτη-μέλη. Λοιπόν, εξού και το ερώτημα. <clears throat> Τι είναι εκείνο το οποίο παρακόλλησε το να σημειωθεί πρόοδο στο πλαίσιο του διοντολογικού κώδικα για την φορολογία επιχειρήσεων, ώστε να επεκταθεί αυτό το πλαίσιο σε πολλέ άλλε καταχρηστικέ μορφέ ε, φοροανταγωνισμού σε αυτό το επίπεδο. Και τρίτον, τελευταίο, διαβάσαμε σε σχέση με τι ειδήσει ε, πληροφορηθήκαμε στην, ε, και στην Ελβετία και στην ΕΕ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει απάμβληνε τις διαπραγματεύσεις ε, με την Ελβετία, τις ε, κατέστησε πιο ήπιες σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα θέλαμε να μας πείτε αληθεύει αυτό και αν αυτό πραγματικά συμβαίνει, τότε γιατί, για ποιο λόγο διότι οι εταιρείε σε σχέση με την Ελβετία το να μην συνεργάζονται και να μην εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο δημιουργεί ζημιά. Και γι' αυτό θα ήθελα να με πληροφορήσετε. Ευχαριστώ. Thank you for your which you Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θετική αξιολόγηση της έτρετους μου εργασίας. Όσον αφορά τα ερωτήματά σας, ή μάλλον καλύτερα τα σχόλιά σας. Συμφωνώ μαζί σας ότι η σημασία της επάταξης της φοροδιαφυγής θα αποκτήσει ακόμα, θα, θα, θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο. Η συγκεκριμένη σας ερώτηση όσον αφορά τον ανταγωνισμό, ε, τον φορολογικό ανταγωνισμό, ναι, όντως αυτό μπορεί να έχει άσχημες επιπτώσεις, αλλά υπάρχει και η ομάδα δεοντολογίας για τα θέματα αυτά και νομίζω ότι μέχρι τώρα ήταν αρκετά επιτυχής η εργασία τους. Όσον αφορά την αυτόματη ή κατόπιν αιτήματο ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτόματη ανταλλαγή. Αλλά όσον αφορά τη saving taxation, ε, την οδηγία αυτή, υπάρχουν τρεις ε, χώρες μέλη που δεν θα συμφωνήσουν εκτός και αν προβληθεί και ο άλλος τρόπος ανταλλαγής ε, ε, πληροφοριών, δηλαδή ο εναλλακτικό μάλλον προς την ανταλλαγή πληροφοριών, δηλαδή και η παρακράτηση. Τώρα υπάρχουν πέντε ευρωπαϊκές χώρες και τα δέκα συνδεδεμένα υπερπόντια διαμερίσματα ε, που έχουν ήδη ε, αναγγείλει αλλαγές όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών του συστήματος, δηλαδή που ισχύει για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, όμως δεν πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή τουλάχιστον μέχρι το τέλος της θητείας μου ενδεχομένως σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων ενδεχομένως σε άτυπο επίπεδο να προχωρήσουμε, αλλά σίγουρα δεν θα ολοκληρωθεί επισήμως η διαδικασία. Το πρώτο βήμα έγινε από την ε, ε, οδηγία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και βεβαίως το να γίνεται λόγος για το τραπεζικό απόρριτο σαν ένα από τα κεντρικά στοιχεία πάταξης της φοροαπάτης, μα αυτό αναφέρεται ήδη στην οδηγία που ανέφερα προηγουμένως. Εκεί γίνεται συγκεκριμένο λόγος για την άρση του τραπεζικού απορρίτου. Επομένως γίνανε τα πρώτα βήματα, απλώς θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή, να προχωρήσει δηλαδή η διαδικασία αυτή. Α, ναι, όσον αφορά την Ελβετία, με ρωτήσατε. Ναι, ναι, έχουμε μπει σε διαδικασίε. Ξεκίνησαν μόλι οι ε, διαδικασίε. Δόθηκε δηλαδή η σχετική εντολή από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Έχουμε ξεκινήσει και με το Λίχτενστάιν, όπω είπα προηγουμένω, και έχουμε ξεκινήσει και με την Ελβετική Συνομοσπονδία. Ευχαριστώ. Για την ΓΚΟΕ, ποιο θα μιλήσει? εσεί μάλιστα, έχετε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την ενημέρωση. Επειδή όπως είπε και ο ίδιος είναι απερχόμενος Επίτροπος, η τοποθέτησή του είχε ένα χαρακτήρα απολογισμού. Ένα γενικόλογο θα έλεγα χαρακτήρα. Ας μου επιτρέψει λοιπόν δύο-τρεις ερωτήσεις γενικού ενδεχομένως χαρακτήρα. Με ενδιαφέρον θα, θα ακούσω τις απαντήσεις του σε ορισμένα θέματα που μας αφορούν και ομολογώ έχει και πολιτικό χαρακτήρα, έχουν και πολιτικό χαρακτήρα ερωτήσει. Το πρώτο, είπατε πολύ σωστά κύριε Επίτροπε ότι μια σωστή και δίκαιη φορολογική πολιτική είναι ένα καλό εργαλείο για να αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη και η απασχόληση. Σήμερα λοιπόν που ζούμε σε πολύ χαμηλούς έως μηδονικούς αριθμούς ανάπτυξης και το πρόβλημα της ανεργίας ανεβαίνει στην Ευρώπη, τι θα λέγατε, πώς θα μπορούσε μια διαφορετική φορολογική πολιτική πράγματι να έπαιζε το έργο, το ρόλο αυτού του εργαλείου. Υπό ποιε προποθέσει επομένω αυτό που σωστά διαπιστώνεται, μια φορολογική πολιτική μπορεί να υποβοηθήσει και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τη απασχόληση, μπορούμε να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο. Η δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στο φαινόμενο της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, το οποίο αν σημείωσα καλά φτάνει στο ύψος ή και ξεπερνάει δύο φορές το ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το ερώτημα είναι, <clears throat> έχετε εικόνα της ακτινογραφίας αυτών που αποφεύγουν να είναι εντάξει στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή, ποιες κοινωνικές ομάδες καταφέρουν να ξεφεύγουν από αυτές τις υποχρεώσεις. Για να σας βοηθήσω στη χώρα μου στην Ελλάδα, αυτές που δεν είναι εντάξει με τις φορολογικές υποχρεώσεις γενικώ είναι οι μεγάλε επιχειρήσει. Επομένω, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να μειωθεί αυτό το φαινόμενο. Προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούν οι έλεγχοι. Και το τρίτο πιο επιμέρους θέμα. Ε, είχα ρωτήσει και τον, και ε, ε, Υπουργό Οικονομικών και τη Σουηδική Προεδρία. Υπάρχει ένα θέμα, το θέμα των offshore εταιριών. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, πού βρισκόμαστε. Γενικώ αξιοποιείται Ω ένα τρόπο αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων. Τι λέτε από αυτού, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει για να περιοριστεί και αυτό το φαινόμενο. Σα ευχαριστώ πολύ. Η φορολογική πολιτική μπορεί να προωθήσει την απασχόληση με δύο τρόπους τουλάχιστον. Πρώτον, η ε, εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά με έντονη εργασία και το λέω αυτό γιατί ε, η μείωση του φόρου προσθέμενης αξίας στις τοπικά παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα οδηγήσει σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό επιμένω στις υπηρεσίες αυτές. Αρχικά, οκτώ κράτη-μέλη άρχισαν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή των μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ για τις υπηρεσίες έντονης εργασίας στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στόχος να δημιουργηθεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι αρχικό του στόχος. Βέβαια, αν αναλύσουμε τα πράγματα σωστά, βλέπουμε ότι δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσει εργασία. Όμω, μετά από μερικά χρόνια, αυτά τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ ήταν τόσο καλά ριζωμένα στα συστήματα κοστολόγησης των χωρών αυτών που οι χώρες αυτές αποφάσισαν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού και μάλιστα προσχώρησαν στο σύστημα αυτό και άλλες χώρες γιατί συνειδητοποίησαν ότι οποιαδήποτε αύξηση των ποσοστών φόρου προσθέμενης αξίας θα δημιουργούσε σε απώλεια θέσεων εργασίας. Επομένως ήταν πολύ σημαντικό για μας να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό και να το καταστήσουμε μόνιμο προκειμένου να αποφύγουμε το να κλείσουν πάρα πολλέ μικρέ και μεσές επιχειρήσει και να χαθούν πάρα πολλέ θέσει εργασίες. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό ο σχετισμός, μολονότι η σχέση είναι κάπω περιορισμένη. Ο άλλο λόγο βέβαια που δεν αποτελεί κοινωνική αρμοδιότητα είναι να συμβουλεύσουμε τα κράτη-μέλη να μειώσουν το φορολογικό βάρος της εργασίας όσον αφορά τις επιδόσεις. Προκειμένου όμως να διατηρηθεί μια καλή ισορροπία στον προπολογισμό και να αυξηθούν οι φόροι για τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού και για την κατανάλωση και να αυξηθούν οι φόροι για τις ε, ζημιές που γίνονται στο περιβάλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την πολιτική απασχόλησης. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Για όσου θεωρούν ότι δεν ακολουθώ σωστά το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να σα πω ότι ο Επίτροπο μπορεί να μείνει λίγο παραπάνω. Επομένω, θα καταφέρουμε να καλύψουμε όλε τι ερωτήσει. Κάναμε ένα πρώτο γύρο από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και θα ήθελα τώρα ή δυνατόν στις επόμενες παρεμβάσεις σας να είστε λίγο πιο σύντομοι γιατί θα χρειαστεί κύριε Επίτροπε να απαντήσετε σε πολύ περισσότερου ε, ευρωβουλευτέ στη συνέχεια. Θα διαβάσω τώρα τα ονόματα με τη σειρά που θα πάρετε το λόγο. Η ακόλουθη. Αυτή είναι η πρώτη τρία, η επόμενη τρεις. Και στη συνέχεια η τρίτη ομάδα. Αν υπάρχει κανεί άλλο που θέλει να πάρει το λόγο, ή που ξέχασε να φέρω το όνομά του, παρακαλώ πολύ πείτε το μου. Εφορτικά δίνω κατευθείαν το λόγο στην Ελίν. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομη προκειμένου να καταφέρουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε και να ευχαριστήσω επίσης και τους συνεργάτες σας από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά στο παρελθόν. Ξέρω ότι ε, το ζήτημα της ε, φορολογικής πολιτικής το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Αναφερθήκαμε επίσης σε διάφορα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε στο Isle of Man, στο Βέλγιο, την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φαίνεται ότι υπάρχουν πολλέ χώρε οι οποίε θέλουν να υιοθετήσουν και τι συστάσει που γίνονται από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να έχουμε τέτοια ανταλλαγή πληροφοριών με την Αυστρία και το Λουξεμβούργο, με συγχωρείτε. Θεωρώ ότι ε, οι χώρε αυτέ δεν έχουν ε, συμμορφωθεί απαραίτητα, ιδίω ε, η Αυστρία με την απέτηση αυτή. Επομένω, α μην εστιαζόμαστε μόνο στι τρίτε χώρε, αλλά α δούμε και τα του μα. Επίση, το ρόλο που θα πρέπει να διδραματίσουν ε, οι ε, ρυθμιστικές αρχές των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αν δεν ε, κάνω λάθος, έγινε αναφορά πρόσφατα και στη χρησιμοποίηση ενός φόρου το BIN και το G20 αναφέρθηκε σε ένα διεθνές πλαίσιο ρύθμιση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενός φόρου για τις υπηρεσίες αυτές. Πιστεύετε εσείς ότι είναι ευκταίο κάτι τέτοιο, δηλαδή να να καταβάλουν περισσότερα ποσά και οι, ίδιες, οι, οι ίδιοι οργανισμοί χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί χρηματικά η κρίση και να μην καταβάλουν τελικά το αντίτιμο μόνο οι φορολογούμενοι. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι το δυνατόν συντομότερη. Τα πιο σημαντικά νομίζω ήδη καλύφθηκαν, προαναφέρθηκαν. Πρόκειται, πρόκειται πρώτα για την εργασία, για την ε, παροχή υπηρεσιών και το μειωμένο ΦΠΑ ε, για τις υπηρεσίες. Ε. Εδώ θα πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ. Αν κατάλαβα καλά, Επίτροπε, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει μια σαφής τοποθέτηση για το πώς ήταν χρήσιμο αυτό ή όχι και το πόσες θέσεις απασχόλησης από αυτά, αυτό το μέτρο δημιουργήθηκαν. Σας κατάλαβα σωστά. Πραγματικά δεν υπάρχει ακόμα τελεσίδικη θέση από πλευρά σας αν αυτό έδειξε ότι είναι υποφελές ή όχι. Δεν έχετε μια οριστική, καθοριστική άποψη για τη μείωση του ΦΠΑ. Δεύτερον, πρόκειται για την καταπολέμηση των φορολογικών οάσεων. Σε σχέση με την φοροεισφορά και την απάτη και τη φοροδιαφυγή αναφέρατε δεν αναφέρατε συγγνώμη, συγκεκριμένα ποσά ως αριθμητικά μεγέθη. Έχετε κάποιες εκτιμήσεις ποιο είναι το ύψος αυτών των ποσών που περνάνε στις φορολογικές οάσεις και εκφεύγουν, διαφεύγουν φορολογίας και κατά τα άλλα. Τι θεωρείτε για τη μείωση του ΦΠΑ ως μέσο για την αναζωογόνηση της οικονομίας. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό, για το μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ για την αναζωογόνηση της οικονομίας. Δεύτερον, για μια στρατηγική διαφυγής ή διεξόδου από την κρίση, exit strategy. Τι θα προτείνατε στα κράτη-μέλη, μέχρι πότε πρέπει να υιοθετηθεί μια τέτοια πολιτική. Ευχαριστώ. Τρεις θα παίρνουμε. Στη συνέχεια Όλε Σμιτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Επίτροπο Νομίζω κάνατε ό,τι περνούσε από το χέρι σας, ό,τι ήταν εφικτό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πεδίο, δυσχερές εγχείρημα, ναρκοθετημένο από παντού. Και ιδιαίτερα το ότι καταφέρατε σε σχέση με τα audiobooks να υπάρχει ένα χαμηλότερο ποσοστό ΦΠΑ, πιο ευνοϊκό, είναι σημαντικό. Το καταφέρατε αυτό. Ακόμα και με λιγότερο πρόθυμους υπουργούς οικονομικών το πετύχατε. Συγχαρητήρια σας ευχαριστούμε. Διαρωτώ με, τι θα έπρεπε να κάνουμε για να καταφέρουμε περισσότερα σε σχέση με αυτά. Εδώ και δέκα χρόνια εμπλέκομαι σε αυτή την προσπάθεια και την παρακολουθώ. Μπορούμε να κάνουμε λόγο για επιβλαβή φοροανταγωνισμό αλλά και για υποφελή φοροανταγωνισμό. Εγώ είμαι υπέρ ενός είδους ανταγωνισμού, ενός θεσμικού ανταγωνισμού ας το πω έτσι. Νομίζω μπορώ να το πω αυτό, είναι θεμητό να το πω. Έχει υψηλότερους φόρους ε, η Δανία. Βρισκόμαστε στην ε, ομάδα των πρωταθλητών αυτών. Παρότι προσπαθούμε να μειώσουμε τους φόρους και τα ποσοστά τους, Πραγματικά όμως πιστεύω ότι θέματα διασυνοριακά που αφορούν το ενόπνευμα, τα ενοπνεύματα, τα τσιγάρα λοιπά, <clears throat> θα πρέπει να δούμε ότι μια ξεχωριστή πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί εδώ έχουμε μεγάλη διασυνοριακή αν θέλετε διακίνηση και λαθρεμπόριο εινοπνευματοδών και σιγαρέτων. Αν θέλετε να αφήσετε κάτι στο γραφείο του επόμενου επιτρόπου, όποιος και να είναι αυτό, αφήστε τουλάχιστον ένα μικρό σύντομο σημείωμα για αυτή την υπόθεση, για την καταπολέμηση αυτού, γιατί αυτό είναι πραγματικά επιβλαβή φοροανταγωνισμό. Σα ευχαριστώ για ό,τι κάνατε. Είμαι ευγνώμων εξετάζοντας την πρώτη ερώτηση από τους τρεις προλαλήσαντες. Ναι, το Βέλγιο άλλαξε την πολιτική του όσον αφορά την ανταλλαγή αυτόματα πληροφοριακών στοιχείων, όσον αφορά εκείνα τα μέρη που έχουν επενδύσεις ε, και ως φορολογικές οάσεις. Γνωρίζω ότι υπήρξε κάποια κινητοποίηση στην Αυστρία, αλλά απέτυχε στο Κοινοβούλιο της Αυστρίας απέτυχε στο ε, Αυστριακό Κοινοβούλιο. Δεν έχω κάποια λοιπόν πληροφορία για κάποιους που θα ήθελαν να ενταχθούν στην λέσχη εκείνων που εφαρμόζουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα με την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι κατά της οδηγίας ε, για τις αποταμιεύσεις ε. είναι ένα είδος μόνο παράτασης που ολοκληρώνεται, εκπνέει αυτή η παράταση. Και όταν το ποσοστό του withholding tax θα αυξηθεί όσον αφορά το 2011 σε 35% ε, τότε θα αλλάξει σίγουρα η κατάσταση άρδιν. Θα δημιουργηθεί ξαφνικά πίεση σε αυτές τις δύο χώρες να αλλάξουν τη θέση τους διότι 35% παρακράτησης φόρου withholding tax δεν θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο μέτρο για α, εκείνους ε, που έχουν ε, αποταμιεύσει στις τράπεζες. Τώρα, όσον αφορά τον φόρο Tobin ή τον φόρο των ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, Νομίζω λογικό ακούγεται, αλλά με βάση την πενταετή μου αυτή πείρα ως ε, επίτροπος ε, για τα θέματα αυτά ε, και τα σχετικά με τη φορολογία, δεν πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορούσε ομοφωνία να επιτευχθεί για το τι χρειάζεται να κάνουμε. Ελπίζω ότι ο επόμενος επίτροπος και για θέματα φορολογίας θα μπορέσει να επομιστεί και να δώσει συνέχεια. Είναι μια λογική προσπάθεια. Αν στεφτεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα όμως από πλευρά του ή όχι, δεν μπορώ να προδικάσω και να πω. Ε, τώρα θα μιλήσω ουγγρικά σε εσά ε, για την ερώτηση που κάνατε πιο πριν και γι' αυτό θα μιλήσω και θα σας απαντήσω στα ουγγρι... ουγγαρέζικα. Τώρα, όσον αφορά την μείωση, το μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ, προσέξτε, το όφελος δεν καταδείχθηκε με κάθε σαφήνεια σε αυτή την περίπτωση. Συμβαίνει αυτό. Τώρα, το 1998, όταν ξεκίνησε μια προσπάθεια διετούς διάρκειας, αυτή η προσπάθεια παρατηνόταν μετά στη συνέχεια και επεκτηνόταν. Και όταν κατέληξα εγώ στο αξίωμά μου 2004, τέλη 2004, τότε αυτή η σκέψη, είχε, αυτή η πρωτοβουλία είχε μακρά προϊστορία. Υπήρχαν δύο δυνατότητες. Ή να τερματιστεί αυτό το σύστημα ή να ανοίξει τελείως. Τώρα το ότι συμμετείχαν οκτώ κράτη μόνο δεν έβαινε καλώς, δεν ήταν εντάξει. Είπα και κατέβαλα προσπάθεια να ανοίξουμε το σύστημα και το καταφέραμε αυτό, το πετύχαμε το 2006. Δέκα επιπλέον χώρες εντάχθηκαν και είπα με, ε, το, σύστημα, με το σύστημα αυτό θα γίνει προσπάθεια ακόμα παραπέρα πέρα να το επεκτείνουμε και να το ανοίξουμε και θα έπρεπε να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα ως διορία για να το πετύχουμε. Βρήκαμε μια λύση, ο πίνακας ο κατάλογος δεν μπορούσε να επεκταθεί απεριόριστα και ακριβώς στο τέλος δημιουργήθηκαν προβλήματα και ήταν ας το πω έτσι βρασιπρόθεσμα μια επιτυχία, εντάξει ανοίξαμε το σύστημα, 18 κράτη συμμετείχαν, όλα τα κράτη που ήθελαν να συμμετάσχουν μπορούσαν και μπόρεσαν να συμμετάσχουν και να προσθεθούν σε αυτό τον κατάλογο. Αλλά εδώ προστέθηκε και ο κίνδυνος. Αν δεν βρίσκαμε μια τελεσίδικη καθοριστική λύση, τότε θα έπρεπε να επανέλθουμε στα, στα στάνταρ ποσοστά και θα καταλήγαμε στα 18 κράτη και αυτό θα ήταν αρνητικό, καταστροφή λόγω θέσεων, απολία θέσεων απασχόλησης. Και γι' αυτό παρακάλεσα τον κύριο Μπαρόζο, Μπαρόζο στη συνέχεια, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη σύνοδο της ΕΕ συγκεκριμένα να αναφέρει αυτή την ιδέα αν δεν εξευρισκόταν μια λύση από πλευρά ΕΚΟΦΗΝ. Και θα έπρεπε να συναχθούν οι συνέπειε, τα συμπεράσματα στη συνέχεια. Διότι σκέφτηκα και είπα ότι μπορεί να μην τα γνώριζαν αυτά οι αρχηγοί κρατών μελών και κυβερνήσεων. Ο κύριο Μπαρόζο το έκανε αυτό και καταλήξαμε ε, σε ένα συμπέρασμα. Ζητήθηκε από το ΕΚΟΦΗΝ να επιλύσει το θέμα μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Καταλήξαμε και σε αυτό. Ήταν το συγκεκριμένο χειροπιαστό αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτή τη προσπάθεια Τώρα όσον αφορά την φορομείωση, φορολογική μείωση ποσοστών ΦΠΑ για την αναζωογόνηση της, οικονομία, αυτό εξαρτάται από τη δράση και από το κράτο, ανακράτο. Είναι σαφέ όταν υπάρχει ένα κράτο όπου είναι υψηλότατο το, δημόσιο το δημοσιονομικό έλλειμμα, τότε σίγουρα είναι ένα επικίνδυνο εγχείρημα να μειώνει κανεί τα ποσοστά φορολογία, διότι το έλλειμμα μεγαλώνει, αυξάνεται. Υπάρχει μεγαλύτερη χρέωση υπερχρέωση, καταλήγουμε σε υπερχρέωση και πρέπει και περισσότεροι τόκοι να καταβάλλονται από πλευρά ενό τέτοιου κράτου. Φαίνεται ίσω προσωρινά να είναι μια τέτοια λύση καλή, αλλά μακροπρόθεσμα συσσωρεύονται προβλήματα και γίνεται προβληματική ε, ε αυτή η κατάσταση. Επιπλέον υπάρχουν επιχειρήματα σε σχέση με την μείωση της φορολογίας. Καλύτερα να συνεχίσει η καταβολή φόρων, αλλά όχι αμέσως το επόμενο, τον επόμενο μήνα ή το επόμενο έτος, αλλά μετά από δύο-τρία χρόνια. Ε, αν όμως ένα κράτος έχει υψηλότατη χρέωση, υψηλά ε, ποσά ε, και είναι χρεωμένο, δεν μπορεί να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία. Τώρα, τι γίνεται με τις φοροάσεις, ε, ποιες είναι οι απώλειες λόγω της ύπαρξης των φορολογικών οάσεων. Δεν μπορεί κανείς να το εκτιμήσει. Είναι 200-253 ε, και όσον αφορά ΦΠΑ περίπου 70 ίσως 3. αυτό είναι μια απλή εκτίμηση και ίσως μπορεί να αληθεύει το ποσό. Υπάρχουν τρεις μεγαλύτερες ομάδες ε, όσον αφορά εινοπνευματόδη ποτά, όσον αφορά τα σιγαρέτα και τα καύσιμα ε, σε σχέση με την δική μου πείρα αυτό δείχνει ότι συμβαίνει. Το πρώτο επιχείρημα όταν υπέβαλε προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξηθεί το ελάχιστο ποσοστό των ειδικών φόρων κατανάλωσης είχαμε το θέμα της επανεκτίμησης. Θυμάμαι όταν παρουσιάστηκε η πρώτη πρόταση για να αυξηθεί το ειδικό καθεστώς έκτακτων δασμών σε σχέση με τα ε, ποσοστά θέλαμε να υπάρξει επανεξέταση διότι 32% ε, ε, από το 1979, από το 92, από το 1992 τα νέα κράτη-μέλη τι έκαναν. Ήταν λογικό ότι επιχειρηματολογούσαν λέγοντας τι θα κάνουμε με το ποσοστό του πληθωρισμού που από το 1992 ήταν πάρα πολύ πιεστικό. Άλλες χώρες βρήκαν απαράδεκτο την αύξηση των ειδικών ε, δασμών και φόρων κατά, στο 32% για τα υνοπνευματόδη Βρήκαμε μια, ένα συμβιβασμό. Ξεκινήσαμε από μια διαφορετική ε, εναλλακτική λύση ως αφετηρία. Είπαμε, και αυτό έγινε το 2004, η ημερομηνία της μεγάλης διεύρυνσης, της μεγάλης έκρηξης Big Bang, όταν τα πολλά τα νέα κράτη-μέλη της Κεντροανατολικής Ευρώπης εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την αφετηρία είχαμε αύξηση 4,5%. Και αυτή ήταν η βάση με την οποία καταφέραμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε αυτήν, αλλά υπήρξε δικαίωμα άρνηση κυρίας λόγω του ζήθου της μπύρας από την τσεχική, τη δημοκρατία της Τσεχίας και επειδή σε σχέση με την επίπτωση για την τιμή της μπύρας δεν θα είχε επίπτωση διότι ήταν υψηλότερο το ποσοστό από την προτινόμενη αύξηση Παρό, παρόλα αυτά όμως ήταν θέμα αρχής για την δημοκρατία της Τσεχίας και έπρεπε να το δεχθούμε αυτό δεν ήταν έτοιμοι να δώσουν το πράσινο φως και να συμφωνήσουν σε αυτή την πρόταση και έτσι με το βέτο απέτυχε εκεί βρισκόμαστε τώρα και το αφήνω αυτό στον διάδοχό μου αν όμως η θέση της Τσεχίας είναι πιο ευέλικτη και έχουμε κάποια μηνύματα ότι θα μπορούσε να ήταν πιο ευέλικτη, θα μπορούσαμε να ε, πετύχουμε αυτή τη συμφωνία. Εκείνο το οποίο βίωσα εγώ είναι ότι για το θέμα αυτής της επαναξιολόγησης, revalorization, υπάρχει αυτό το δεδομένο επιχείρημα, αλλά υπάρχουν και άλλα πιο λογικά, πιο αποδεκτά επιχειρήματα και στην περίπτωση των ε, σιγαρέτων και των ενοπνευματοδών ποτών έχουμε και τα θέματα υγείας και τις επιπτώσεις εις βάρος της υγείας. Στην περίπτωση των ε, καυσίμων είναι η βλαπτική επίδραση στο περιβάλλον, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Όταν γίνεται λόγος λοιπόν για τον, την αύξηση της ειδικής φορολόγησης στο ντίζερ για να αποφύγουμε τον τουρισμό εκείνων που περνάνε σύνορα για να γεμίσουν τα ντεπόζιτά τους με ντίζερ, το τελικό αποτέλεσμα ποιο ήταν ότι χιλιάδες επιπλέον μη χιλιόμετρα καλυπτόντουσαν και πάρα πάμπολοι χιλιάδες τόνοι διοξιδίου του άνθρακα εκλειόντουσαν στην ατμόσφαιρα για να κάνουν αυτά τα ταξίδια και να προμηθευτούν αυτό το καύσιμο έναντι για παράδειγμα των φορολογικών ωφελών που θα είχαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπούλμαν, Άλβαρες και κάθε. Κύριε Μπούλμαν. Κύριε Πίτροπε, εσείς στην εισαγωγική σας παρουσίαση αναφέρατε κάτι και είπατε ποιο έργο πρέπει να επιτελεί και μπορεί να επιτελεί η πολιτική για τα θέματα φορολογίας. Όχι μόνο την δίκαια εξισορρόπηση των βαρών και τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και την αλλαγή της βιομηχανικής κοινωνίας και την προσαρμογή της περιβαλλοντικά, οικολογικά και για τον εξυγχρονισμό των βιομηχανικών μας εγκαταστάσεων και όλα αυτά τα βρίσκω αξιόλογα και πραγματικά θετικά το ότι τα προτείνατε. Τώρα, ένα παράδειγμα να δώσω. Στη συζήτηση βρίσκεται το ότι χρειαζόμαστε ένα φόρο ευρωπαϊκό για τα ορυκτά καύσιμα. Δεν θέλω να πω ότι είμαι εναντίον, διότι ακριβώς αυτή η λειτουργία η φορολογική είναι εκείνη που μπορεί να δώσει αποτελέσματα. Όμως υπάρχει σύγκρουση όσον αφορά τα συμφέροντα και τους στόχους. Τα κράτη-μέλη προσπαθούν να μεταθέσουν αυτό στις Βρυξέλλες. Στις χώρες μας έχουμε την ε, αυξημένη επιβάρυνση των καταναλωτών που βρίσκονται σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης. Δεν είναι απλό αυτό. Αν πάμε στο άλλο άκρο της συζήτησης όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αγορές, έχουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση των αντιμαχωμένων. Αν εδώ τώρα οι φόροι βράχοι πρόθεσμα επιβληθούν στους όσους εμπλέκονται στην οικονομία και όσον αφορά και τα κέρδη και σε σχέση με τις εναλλακτικέ επενδύσεις και τα λοιπά, τότε ενισχύουμε ταυτόχρονα την αηφορία στην, στις επενδύσεις την αηφορία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις επενδύσεις διότι αυτές καθιστούν περισσότερο ανταγωνιστικές αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά κερδοσκοπικές τάσεις. Έχει λοιπόν αυτό διτά μια υποφελή δράση. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν και αυτή την πολιτική και πείτε μας την προσωπική σας άποψη γι' αυτό. Μήπως εδώ θα έπρεπε να προχωρήσει το θέμα της διεθνούς φορολόγησης ή της επιβολής ενός φόρου ή τέλους επί των συναλλαγών και να δούμε τι μπορεί να γίνει μακροπρόθεσμα. Να δούμε πώς μπορούμε να ευνοήσουμε τη μακροπρόθεσμη επένδυση έναντι των βράχυπρόθεσμων άμεσων και κοντόθωρων επενδύσεων. Αυτό θα ήθελα να πω και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω εξ ονόματος της ομάδας μας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε ευγνώμονες ότι ποτέ δεν εγκαταλείψατε το θάρρος σας, τις γενναίες σας θέσει να είσαστε υπέρ λογικού συστήματος φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια από τις πιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι τα κράτη-μέλη πάντα εμένουν και επιμένουν στα δικά του συμφέροντα. Γι' αυτό από πλευρά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ και κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Μαντελένα Άλβαρες, uh, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε, διότι πιστεύω ότι είναι πλήρης, ε, περιεκτική η πληροφόρηση και καλά στοχοθετημένη. Σας συγχαίρω για την πρόταση οδηγίας και που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία. Είχα και αναλάβει ρόλο ε, κοινοβουλευτική εκπροσώπου για αυτή την έκθεση και πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρόταση που είναι φιλόδοξη είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει σε αίσιο τέλος και όταν θα μπορέσουμε με, πέρα από διμερεί συμφωνίες ε, να ολοκληρώσουμε αυτές τις πτυχές ε, μεταξύ μας ως κράτη. Υπάρχει κάτι που θέλω να υπογραμμίσω εδώ, διότι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν εδώ ε, να υπάρχει ο συγκερασμός της βούλησης και της θέλησης και της ικανότητας για δράση. Και εδώ έχουμε το θέμα της ηθικής στα θέματα φορολογίας που είναι πολύ σημαντικά για τους πολίτες η βούλησή μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτή την ηθική και για την ε, ικανότητα να δράσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για παράδειγμα ως ε, στοιχείο να μπορέσει να λειτουργήσει. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα κύριε πίτροπε. Η πρώτη όσον αφορά την ε, άρση του απορρίτου, του τραπεζικού απορρίτου. Ποιο εμπόδιο μπορεί να υπάρχει στο Συμβούλιο. Τι θα γίνει σε σχέση με κάποια προσκόμματα ή εμπόδια από πλευρά του Συμβουλίου. Δεύτερον, για την ανταλλαγή πληροφοριών θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα ήταν δυνατόν να είσαστε πιο σαφείς στην τοποθέτησή σας στην ε, ε, παρουσίαση εξέβρεσης λύσης ε, για το πρόβλημα του άρθρου 8. Ευχαριστώ. Um, monsieur Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για την διαφάνεια με την οποία μας μιλήσατε και για την ποιότητα των λεγόμενων σας. Ε, θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα ερώτημα παρόμοιο με το αυτό του κυρίου Μπούλμαν ε, σχετικά πρώτον με τη διάσκεψη κορυφής της ε, Κοπενχάγης. Πλησιάζει και θα ήθελα να ξέρω όσον αφορά την οικολογική φορολόγηση ε, τι κατά την άποψή σας θα πρέπει να γίνει έτσι, έτσι ώστε να προσανατολιστεί ο τρόπος παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε έναν τρόπο πιο συνεκτικό προς την ε, φιλικά διακείμενη προς το περιβάλλον Ένωση. Επίσης, ε, ποια είναι τα σχέδια της επόμενης θητείας της Επιτροπής όσον αφορά αυτά τα θέματα και τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για την Border Tax Adjustment, λέει ο μιλητής στα αγγλικά. Δεύτερο ερώτημα, ε, όσον αφορά τους φορολογικούς παραδείσους. Μας είπατε ότι έχουν προβληθεί κυρώσεις ήδη από την άνοιξη του 2010 ε, για τα, τις χώρες ε, οι οποίες δεν θα συνεργαστούν. Αλλά ε, καταλαβαίνετε ότι ε, διαπιστώνουμε ότι από τη στιγμή που η μη συνεργασία είναι μηδέν, ε, τότε θα έχουμε μηδέν κυρώσεις. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας άλλα κριτήρια αξιολόγησης όσον αφορά τον, τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται και καθορίζεται την μη συνεργάσιμη αρχή και έτσι ώστε οι κυρώσεις να μην μείνουν κενό γράμμα και να είναι πραγματικές κυρώσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω πιο σύντομες απαντήσεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ε, θα υπάρχουν άλλες δύο-τρεις ομάδες ερωτήσεων. Βεβαίως εμείς θέλουμε να δώσουμε κάποιες νέες, κάποιους νέους προσανατολισμούς όσον αφορά την, ε, ε, όσον αφορά κάποιες μορφές ή είδους ε, ή είδη φόρων όπως ας πούμε φόρος για ορεικτά καύσιμα κτλ. Και αυτού του είδους η φορολόγηση δίνει και το στίγμα λίγο της πολιτικής μας ε, και πιστεύουμε ότι η μέχρι τώρα ε, πολιτική και οι μέχρι τώρα αποφάσεις μας ε, είναι λογικές και φαντάζομαι ότι θα γίνουν δεκτές από όλες τις φορολογικές αρχές. Η διοικητική συνεργασία, καθώς επίσης και η άρση του τραπεζικού απορρίτου, είναι, δεν πιστεύω ότι στο Συμβούλιο θα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες αυτές δυσκολίες. Βεβαίως, θα υπάρξουν κράτη-μέλη που δεν θα πούν άμεσα ναι. Ακόμα και όταν παρουσιάσαμε και υποβάλαμε την πρότασή μας, ε, υπήρξαν κάποιες τροπολογίες όσον αφορά ε, την ε, οδηγία. Ε, ε, σχετικά με την οδηγία για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Αλλά μετά όμως τα πράγματα άλλαξαν και ακολουθώντας και την αξιολόγηση αυτής της ε, οδηγίας και την φορολόγηση αποταμίευσης είδαμε ότι χρειάστηκαν ένα-δυο μήνες έτσι ώστε να κερδίσουμε έδαφος και στην εκοφήν που, στο Συμβούλιο Εκοφήν ακολούθησε είχαμε διαφορετικές ε, απόψεις. Επομένως πιστεύω ότι και στην προκείμενη περίπτωση, έστω μετά από συζητήσεις, έστω μετά από κάποιο διάστημα θα επιτύχουμε την άρση του τραπεζικού απορρίτου και θα έχουμε το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Όσον αφορά την πράσινη ε, ε, φορολόγηση, τη διάσκεψη κορυφής Κοπενχάγης, πρέπει να σας πω ότι μελετήσαμε προσεκτικά την ε, γαλλοβρετανική πρόταση σχετικά ε, με διαφοροποιημένα ε, ποσοστά όσον αφορά τα πράσινα προϊόντα και όσον αφορά και τις και όσον αφορά και την μείωση των ποσοστών ε, ΦΠΑ. Όμως μετά από συζήτηση ε, φάνηκε ότι η μείωση των ποσοστών ε, ΦΠΑ δεν είναι ενδεχομένως ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να βοηθήσουμε τα πράσινα προϊόντα. Κάποια επιδότηση ίσως θα ήταν πολύ καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Όντως θα πρέπει να δώσουμε κάποιο πλεονέκτημα στα πράσινα προϊόντα σε σχέση με τα ενεργοβόρα και παραδοσιακά παραδοσιακά προϊόντα. Ε, θα πρέπει να δούμε εάν θα είναι κάποιες εκπτώσεις φόρου, αν θα είναι μειωμένος ΦΠΑ, εάν θα είναι άμεση ε, επιδότηση. Οπωσδήποτε θα πρέπει να επιλέξει η Επιτροπή ανάμεσα από θέματα επί των οποίων θα έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη και προτάσεων που θα έχουν ε, συμφωνήσει. Τώρα, πιστεύω ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση Κατά την ε, άποψή μου ε, θα πρέπει όσον αφορά τα πράσινα προϊόντα να προχωρήσουμε στην ε, οδό που έχουμε ήδη ξεκινήσει της εμπορίας των εκπομπών καθώς επίσης και μιας πιο, γενικευμένης, πιο γενικευμένου φόρου για, τον, για το διοξίδιο του άνθρακος. Το πραγματικό ερώτημα είναι οι χώρες ε, οι οποίες έχουν ανανεώσει τις ε, δεσμεύσεις τους ε, μετά από την ανακοίνωση του προγράμματος Επιτροπής 2001-2010 και που δεν έχουν βελτιώσει καθόλου τις επιδόσεις τους, τότε εκεί θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις έτσι ώστε οι χώρες αυτές να αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους. Έχουμε, λέει η Πρόεδρος, άλλους πέντε ομιλητές ε, και θα δώσω το λόγο και στους πέντε και δίνω μάλιστα ταυτόχρονα και περισσότερο χαρτί στον Επίτροπο γιατί θα έχει πολλές ε, ερωτήσεις για να απαντήσει. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και για την παρουσία σας, για την εργασία σας αλλά και την υπομονή σας. Ε, θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Κλίνς προηγουμένως, δηλαδή με την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ε, στην ε, Γαλλία υποτίθεται ότι θα, υπήρξε, θα υπήρχε ταυτόχρονα μείωση των τιμών. Αλλά μετά από τρία δις που δαπανήθηκαν για το μέτρο αυτό ακόμα περιμένουμε τη μείωση των τιμών. Ε, σας, ρωτώ, λοιπόν, σας ζητώ λοιπόν να αφήσετε ένα πραγματικό μήνυμα, όχι τεχνοκρατικό μήνυμα στον διάδοχό σας, στον αντικαταστάτη σας ε, περάσαμε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Ε, οι χώρες μας έχουν πλέον τεράστια ελλείμματα, γνωρίζουμε τα προβλήματα ε, και γνωρίζουμε επίσης ότι βεβαίως μπορεί να υπάρξει και πρέπει να υπάρξει ενδεχομένως κάποια, κάποιος ανταγωνισμός όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα, αλλά σαφέστατα όχι ένας ανταγωνισμός ο οποίος θα καταλήξει σε κούρσα η οποία τελικά θα έχει έχει αρνητική έκβαση για τους πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε εκλεγεί από τους ε, πολίτες μας ε, και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε μερικά πράγματα. Ε, είναι γεγονός ότι μπορούν και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ζυμώσεις αλλά όχι τέτοιες που θα οδηγήσουν τους πολίτες στο συμπέρασμα ότι δεν ανήκουν τελικά σε ένα σύνολο ε, στο οποίο επικρατούν όροι ευγενούς άμυλας ε, κτλ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσετε ένα κληροδότημα που θα αφορά το σύνολο των πολιτών και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σκούτας, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στα πλαίσια της κρίσης η απάντηση που δώσαν τα κράτη-μέλη ήταν διαφορετική. Κάποια κράτη αποφάσισαν να αυξήσουν τη φορολογία ή επινόησαν και νέους φόρους. Κάποια άλλα κράτη-μέλη αποφάσισαν να μειώσουν τους φόρους, να καταργήσουν κάποιους φόρους. Ποια είναι η αποψή σα σε σχέση με αυτό, δηλαδή ποια, ποια κράτη απάντησαν καλύτερα στην κρίση. Και στα πλαίσια της κρίσης αυτής, ξέρω ότι στην ημερήσια διάταξη του G20 θα προτινόταν ε, ένας γενικός φόρος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενιαίος φόρος. Ποια είναι η άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ. Ναι κύριε Κόβατς. Ουσιαστικά δύο σύντομες ερωτήσεις έχω μόνο. Τόμπιν Στόιερ και τέλος συναλλαγών αρκετές φορές αναφέρθηκαν σήμερα. Έχω μια επικαιροποιημένη έκδοση της ε, επιστημονικής υπηρεσίας ε, της ε, Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής. Η επιστημονική υπηρεσία του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Κοινοβουλίου ερμηνεύει τη συνθήκη της Λισαβόνας με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιες μορφές φορολόγησης δεν είναι πλέον εφικτές και αναφέρεται στα άρθρα 63 και 65 της συνθήκης Λισαβόνας. Η Τη συνθήκη ε, για την λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και λέει τέτοιου είδου φόροι δεν είναι επιτρεπτοί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν και με τη συνθήκη τη Λισαβόνα ε, διευθετείται τελεσίδικα πλέον αυτό το θέμα. Πώ το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε με αυτήν την άποψη. Είναι μια μονομερή ε, γερμανική ερμηνεία αυτή. Η δεύτερη οδηγία αφορά την ερώτηση αφορά την οδηγία 2008 του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου για τον, τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών από την επιστημονική υπηρεσία του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου ερμηνεύεται ότι εκεί που υπάρχει αυτό το ποσοστό φορολόγηση ε, κύκλου εργασιών μπορεί να διατηρηθεί στι χώρε που υπάρχει, αλλά άλλε χώρε δεν μπορούν να το εισαγάγουν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, ε, με την πίεση που υπάρχει κάποιε χώρε που είχαν αυτό το ποσοστό μπορούν τώρα να το να υπαναχωρήσουν και να μην λειτουργήσει πια. Πώ το κρίνετε αυτό εσεί, ευχαριστώ. Περβόν σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ζωή σας μπορώ να πω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε κάπως δύσκολα αλλά τελειώνει με επιτυχία. Είναι άραγε η, ε, το σύστημα ομοφωνίας το Συμβούλιο και η αντίδραση των κρατών μελών που μας έκανε τελικά να έρθουμε τόσο κοντά. Βοήθησε αυτό την καλή συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όποια και να είναι η απάντηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Πρώτο, μειωμένα ποσοστά φόρου προστιθέμενης αξίας. Όσοι πιστεύανε ότι έπρεπε να διονυστεί το σύστημα μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ γιατί είχε συνεσφέρει πολύ θετικά τελικά και γιατί ε, ουσιαστικά είχε να κάνει κυρίως με τις υπηρεσίες έντονης εργασίας, είχαν τελικά δίκιο. Εγώ όμως θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα καταστρεπτικές οι πολιτικές αυτές υποσχέσεις, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση του φόρου προσθέμενης αξίας για τα εστιατόρια, με πραγματικές επιπτώσεις πολύ διαφορετικές από αυτές που μας είχαν πει οι δήμονες του τομέα. Αυτές λοιπόν τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες θα ήθελα να τις καταγγείλω. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν στα πλαίσια της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γίνει μια κάποια μελέτη αντικτύπου όπως ήθιστε να λέγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, πραγματικότητα της κατάστασης, για τις πραγματικές δηλαδή επιπτώσεις των μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ που έχουν πλέον παγιωθεί τόσο για τις υπηρεσίες έντονης εργασίες όπου αποδείχτηκε ότι αυτά τα ποσοστά, τα μειωμένα ποσοστά ήταν χρήσιμα και ότι τελικά κατέδειξαν ότι μπορούν να νομιμοποιηθούν εργασίες, θέσεις εργασίας που στο παρελθόν ήταν στην μαύρη αγορά παράνομες. Από την άλλη όμως μήπως θα έπρεπε να γίνει και μια μελέτη αντικτύπου για να δούμε τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις που είχαν τα μειωμένα ποσοστά φόρου προσθέμενης αξίας στα εστιατόρια που δεν επωφελήθηκε καθόλου ο καταναλωτής και όπου ουσιαστικά εδώ πέρα η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική από τις αρχικές υποσχέσεις που είχαν δοθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε έναν προκάτοχό σας που είχε πολύ καλές και αυτό σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφερθώ στον Μάριο Μόντι, ο οποίος είχε αναφερθεί σε ζητήματα φορολογικά και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στιγμή καμπής αν θέλετε. Θα μπορούσαμε να αναφερόμασταν όπως στο παρελθόν στη μεγάλη αυτή κοινή αγορά χωρίς να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες στις λειτουργίες της αγοράς αυτής. Και δεν ξέρω πώς θα σχετιζόταν, αν θέλει, την προσέγγιση αυτή μια ενιαία εσωτερική αγοράς με τις προτάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν για ένα ενιαίο σύστημα φορολόγησης. Πιστεύετε ότι ε, μπορούμε αυτή τη στιγμή να βρούμε μία διέξοδο στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ε, μία δέσμη μέτρων προκειμένου να προωθηθούν οι προτάσεις τις οποίες μας παρουσιάσατε και να μην μπλοκαριστούν από έναν ε, επίτροπο. Και τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει τις προτάσεις αυτές. Τέλος. Όσον αφορά τον ε, φόρο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα βρίσκανε μια τέτοια πρόταση ιδιαίτερα ελκυστική και εσεί ο ίδιος είπατε για ποιο λόγο θα μπορούσε να θεωρηθεί μια τέτοια πρόταση φορολογήση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ιδιαίτερα ελκυστική. Τι υποδομή όμω χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα, γιατί κάθε φορά που συζητείτε στο παρελθόν αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Θεωρώ ότι το ερώτημα αυτό τίθεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, να δούμε αν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τέτοιο σύστημα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν υπάρχει δηλαδή ένα κοινό πλαίσιο για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα και σε ένα δεύτερο επίπεδο να δούμε αν θα μπορούσε ένα σύστημα τέτοιο κοινοτικό να λειτουργήσει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί το ζήτημα, ενδεχομένω η απάντηση να είναι πολύ εύκολη και να είναι ένα απλό όχι. Νομίζω όμω ότι πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήσει αυτέ, αν θέλουμε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ στην εστίαση. Πολλοί αναφερθήκατε στο ζήτημα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι εξ αρχής ήμουν υπέρ αυτής της πρότασης, δηλαδή της επέκτασης των μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ για τα catering και για τα εστιατόρια. όχι επειδή επέμεινε πάρα πολύ στο ζήτημα αυτό ο πρώην Γάλλος πρόεδρος κατά την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά επειδή θεωρούσα ότι ήταν άδικο σε 11 κράτη-μέλη να ισχύουν, να μπορούν να εφαρμοστούν μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ, πράγμα το οποίο έγινε, ενώ στι υπόλοιπε χώρε ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν τέτοια μειωμένα ποσοστά. Θεώρησα λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανένα λόγο να υπάρχει μια τέτοια διακριτική μεταχείριση, διακριτική αντιμετώπιση των Ευρωπαίων πολιτών από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Όταν ξεκίνησα τη θητεία μου σε 11 χώρε τα μειωμένα αυτά ποσοστά μπορούσαν να εφαρμοστούν ενώ σε 16 άλλε χώρε δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν τέτοια μειωμένα ποσοστά στα εστιατόρια. Θεώρησα λοιπόν ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα κοινό πεδίο δίκαιο για όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιό μου θα πρέπει να λάβει υπόψη του, καταρχάς, την αποστολή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ποιος είναι ο στόχος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με τη συνθήκη της Ρώμης, την εποχή της συνθήκης της Ρώμης θέλαμε να αποφύγουμε έναν επόμενο πόλεμο και μακροχρόνια να καταρρύψουμε τον διαχωρισμό της Ευρώπης που είχε προκύψει με τον ψυχρό πόλεμο. Αυτά ίσχυαν στη συνθήκη της Ρώμης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον τέτοιο διαχωρισμό στην Ευρώπη, δεν υπάρχει τείχος του Βερολίνου, δεν υπάρχει σιδηρού παραπέτασμα, δεν παραμονεύει κάποιος, δεν ροχεύει κάποιος πόλεμος. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δώσουμε καλύτερα επίπεδα ζωής, διαβίωσης, καλύτερα επίπεδα ασφάλειας και καλύτερη περισσότερη ελεγγύη για περίπου 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και, και θα πρέπει να καταστήσουμε, αν θέλετε, τις νέες αυτές συνθήκες διαβίωσης πολύ πιο βιώσιμες. Επομένως, η φορολογική πολιτική θα πρέπει να εξυπηρετεί αυτούς τους γενικούς στόχους, καθώς επίσης και τις βασικές στρατηγικές και τους συγκεκριμένου στόχους που θέτουμε προκειμένου να πετύχουμε του, την, τις πολιτικέ. αυτές πολιτικές. Το επόμενο λοιπόν άτομο που θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιό μου θα πρέπει να λάβει την παράμετρο αυτό, αυτή πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του. Ότι ε, η φορολογική πλέον πολιτική στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους. Συμφωνώ επίσης μαζί σας ότι θα πρέπει να έχουμε δίκαιε συνθήκες ανταγωνισμού όσον αφορά τη φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν θα πρέπει σε κανένα περίπτωση να εγκρίνουμε συνθήκε ανταγωνισμού στην φορολογική πολιτική που θα είναι επιζήμιε για τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ ότι τα κράτη-μέλη δεν αντιμετώπισαν με τα φορολογικά κίνητρα με τον ίδιο τρόπο την χρηματοοικονομική κρίση. Άλλα κράτη-μέλη αύξησαν του φόρου, αλλά πάλι μείωσαν φόρου. Άλλα κράτη-μέλη κατήργησαν φόρου ή επινόησαν νέου φόρου. Δεν υπάρχει σίγουρα μία γενική παγκόσμια συνταγή που θα μπορούσε να ακολουθηθεί. Σε ορισμένε χώρε τα πράγματα είναι όπω ο flat tax, το σύστημα αυτό flat tax, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε κάποια κράτη-μέλη. Και όταν έθεσα το ερώτημα αυτό μου είπαν ότι δεν αποτελεί ο φόρος αυτός κοινοτική αρμοδιότητα. Αν μία χώρα θεωρεί ότι ένα σύστημα φορολόγησης flat tax είναι καλύτερο από ένα προοδευτικό σύστημα, τότε μπορεί να το επιλέξει. Είδα όμως ότι υπήρχαν όλο και περισσότερα κράτη-μέλη, κυρίως νέα κράτη-μέλη, που χρησιμοποιούσαν το σύστημα flat tax και φαίνεται ότι ορισμένες χώρες τώρα επιθυμούν να επιστρέψουν στο προηγούμενο σύστημα, το Progressive Tax System. Δεν υπάρχει σίγουρα λοιπόν ένα κοινό σύστημα που, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν όλες οι χώρες. Αποφασίζουν μεμονωμένα να αυξήσουν ή να μειώσουν φόρους και αυτό έχει να κάνει κυρίως με, με την εθνική οικονομική κατάσταση, με τον εθνικό προπολογισμό. Αν μια χώρα χρειάζεται περισσότερα έσοδα δεν μπορεί να μειώσει τους φόρους. γιατί τότε θα πρέπει να βρει τα απαραίτητα κίνητρα προκειμένου να καταφέρει να κάνει τον πολίτη, τον Ευρωπαίο πολίτη σε κάθε χώρα να καταβάλει περισσότερους φόρους και θα πρέπει όμως παράλληλα ένα τέτοιο μέτρο να μην, εφαρμοστεί άμεσα αλλά να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και στους πολίτες. Τώρα, Οι περισσότεροι επίτροποι θεωρούν ότι ο φόρος για τις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Άλλοι πάλι επίτροποι θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Εφόσον όμως χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει όχι μόνο να μείνει σε κοινοτικό επίπεδο με τέτοια φορολόγηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, αλλά να περάσει και σε παγκόσμιο επίπεδο, μόνο όταν θα λειτουργήσει σωστά. Αυτό όμως καθιστά το όλο εγχείρημα πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο προβληματικό. Όσον αφορά τη μελέτη αντικτύπου, την αξιολόγηση αντικτύπου. Ναι, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια τέτοια μελέτη αντικτύπου από τα διδάγματα τα οποία είχε αποκομίσει από τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ για τις υπηρεσίες έντασης εργασίας, προκειμένου να δούμε αν το σύστημα ήταν σωστό ή όχι. Το 2008 ή το 2009 ήμασταν υποκαθεστώς πίεσης. Έπρεπε να βρούμε μια συμβαστική λύση η οποία θα έπρεπε να μονιμοποιηθεί στη συνέχεια. Γιατί αν δεν βρισκόταν μια τέτοια λύση, 18 χώρες θα έπρεπε να επιστρέψουν στο κλασικό σύστημα ποσοστών ΦΠΑ και αυτό θα ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω, γι' αυτό ακολουθήσαμε τον άλλον δρόμο, των γενικευμένων δηλαδή μειωμένων ποσοστών ΦΠΑ για όλες τις χώρες. Η απάντηση στο τελευταίο σε είναι όντως αρνητική, όντως θα πρέπει να ελέγξουμε περισσότερο αν το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο εκτός μικροφώνου η παρατήρηση της κυρίας Μπερές. Η απάντηση είναι δεν έχω άποψη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω πολύ καλά το δικείμενο δεν έχω διαμορφώσει άποψη. Well, thank you very much, uh, uh, uh, Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. That, that has been quite a, tour de force that you have given. Πραγματικά επιδείξατε ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερο δυναμισμό στην, ε, στις, ε, στο να απαντήσετε αυτές τις πολυπληθείς ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε που μείνατε και αυτή την επιπλέον μισή ώρα. σίγουρα όλοι οι συνάδελφοι, κυρίως δε αυτοί που σας γνωρίζουν και από την προηγούμενη θητεία, σας ευχαριστούν και εύχονται και ευόδοση των εργασιών σας στη συνέχεια να υπενθυμίσω ότι την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έχουμε και μια συνάντηση της Επιτροπής μας. Επιτρέψτε μου, λέει ο κύριος Κόβαξ, να δραθώ της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για την καλή συνεργασία ε, που ε, είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα ήθελα ιδιαίτερος να ευχαριστήσω την Περβάνς Μπερές που ήταν ε, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου, αλλά βεβαίως και την ε, πρόεδρο. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, στα στιβαρά χέρια γυναικών βρίσκεται η οικονομική πολιτική και αυτό είναι πολύ θετικό.